και ευτυχώς ζεστάθηκε λίγο ο καιρός. Αν δεν έχετε αντίρρηση μπορούμε να κάνουμε δεκτή την ημερησία διάταξη. Τα πρακτικά της 22ης και 23ης Ιανουαρίου μπορεί να γίνουν δεκτά επίσης εφόσον δεν έχετε αντιρρήσεις. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις από πλευράς της Προέδρου, οπότε θα ξεκινήσουμε αμέσως Α, έχει ζητήσει ο κύριος Βαντερκάμπ το λόγο. Ένα μικρό... Να προσθέσω ένα μικρό σημείο. Ε, ήσασταν, γίνατε 39 ετών χτες. Εξ ονόματος λοιπόν της Επιτροπής και των μελών της θα ήθελα να σας συγχαρώ. Δεν θα τραγουδήσουμε, αυτό ίσως να το κάνουν στην Επιτροπή Πολιτισμού αλλά παρόλα αυτά θέλουμε να, μας ευχη... να σας ευχηθούμε δύναμη και επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ το σύνολο της Επιτροπής για τις ευχές της. Αλλά είμαι ακόμα λίγο νεότερη από τον κύριο Μακρό. Είμαι λίγο κάτω από 40. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο σημείο, διαδικασία ε, ρύθμισης και ελέγχου για τις ψυχολογικές εξετάσεις του προσωπικού, του υπταμένου προσωπικού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να υπάρχει δυνατότητα προκαταρκτικού ελέγχου. Θέλουμε και εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερωθούμε πλήρως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει το έγγραφό της περαιτέρω. Ελπίζω ότι η συζήτηση σήμερα θα βοηθήσει την κατάσταση και θα προσφέρει στο θέμα αυτό του ψυχολογικού ελέγχου των ψυχολογικών τεστ του υπτάμενου προσωπικού. Μετά από την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ξεκινήσει η συζήτηση. Ο κύριος Ζωακίμ Λουκίν είναι ο υπεύθυνος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Έχετε το λόγο κύριε Λουκίν. Σας ευχαριστώ. Έχω δύο συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την ΑΙΖΑ. Το έγγραφο αυτό στην ουσία είναι κάτι το οποίο ακολουθεί την υπόθεση της ε, γερμανικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους ε, του 15 του ατυχήματος που έγινε τότε ε, εξετάσαμε τις προτάσεις αυτές και κάναμε 11 περαιτέρω προτάσεις έτσι ώστε να υπάρχει σωστή ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για την ψυχολογική υγεία του υπτάμενου προσωπικού. Δημιουργήθηκε επίσης και ε, μια ομάδα task force που αντιπροσωπεύει 14 ε, ε, μεγάλες αεροπορικές επιχειρήσεις εξέτασε τα γερμανικά συμπεράσματα και τον Ιούλιο κατέληξε σε έξι συστάσεις. Η πλειοψηφία των συστάσεων αυτών είχαν καλυφθεί και από την γνωμοδότηση της ESA σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις του υπτάμενου προσωπικού που περιλαμβάνει και μια συνολική ψυχολογική αξιολόγηση τα ιατρικά κέντρα και οι εξεταστές ε, ε, θα πρέπει να καταγγέλουν, να αναφέρουν μάλλον τις ατελείς ιατρικές εξετάσεις. Η τελική διακανονιστική ρύθμιση θα τεθεί σε λειτουργία το 2018. Το νομικό κείμενο το οποίο σας παρουσιάζω σήμερα έχει σαν στόχο να εισάγει επίσης ε, υποχρεωτικούς ελέγχους για τις ναρκωτικές ουσίες και ε, το ενόπνευμα, όπως επίσης και ε, ειδικέ εξετάσεις μετά από προηγούμενη αποτυχία ή μετά από ατύχημα. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα ελεγκτικό το οποίο να δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και να μην δημιουργεί μια ατμόσφαιρα τιμωρητική. Μια άλλη, σύμφωνα με μια άλλη σύσταση, ε, αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο είναι καρπός των συζητήσεων με τους εμπλεκομένους από το 16 και μετά. Οι νομοθετικές προτάσεις βασίζεται στη γνωμοδότηση 14 του 2016 της ΑΕΣΑ και με βάση επίσης την 965 του 12 στην ουσία εδώ παρουσιάζονται προτάσεις βελτίωσης του ε, ελέγχου του ιατρικού του προσωπικού. Συζητήθηκαν και στα πλαίσια τεσσάρων συνεδριάσεων της Διοικητικής Επιτροπής της ΕΑΖΑ και νομίζω ότι τον Φεβρουάριο ε, υιοθετήθηκε το τελικό κείμενο συνενετικά με βάση την 14 του 2016 και θα τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2018. Τώρα, να περάσω στο περιεχόμενο, αν θέλετε, της ε, οδηγίας. Σχετικά τώρα λοιπόν με τους κανόνες που θα εφαρμόζονται από εδώ και πέρα. Δε, πρώτον, προληπτικά μέτρα σαν παράδειγμα ε, ψυχολογικός έλεγχος και αξιολόγηση του προσωπικού του υπτάμενου πριν ξεκινήσουν την ε, πτυτική τους δραστηριότητα. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνεται ε, πριν από την πρώτη εμπορική πτήση. Δεύτερον, θα πρέπει να καθιστούμε ικανούς τους μηχανισμούς ελέγχου να έχουν διάρκεια καθ' όλη την επαγγελματική δραστηριοποίηση των πιλότων ακόμα και της προσωρινής παύσης από την δραστηριότητα αυτή. Επίσης, συστηματικές ε, διαδικασίες ελέγχου σχετικά με κατανάλωση ουσιών και εινοπνευμάτων, υνοπνευματοδών, συγγνώμη, ε, και αυτά όλα θα πρέπει να ολοκληρώνονται πριν από την εναρκτήρια, αν θέλετε, εμπορική τους πτήση. Τα δεύτερα μέτρα τώρα είναι διορθωτικά μέτρα σχετικά με, τον, τα αλκοτέστ, το σύστημα το οποίο προβλέπετε εξελίσσεται σε διαφορετικές ε, ε, ευκαιρίες. Πρώτον μετά από ένα σοβαρό ατύχημα, μετά από ένα απλό ατύχημα, μετά από έλογες υποψίες και μετά επίσης από επιστροφή που ακολουθεί την διακοπή της δραστηριότητας της πληκτικής. Επίσης θα γίνονται και έλεγχοι ε, ράμπας όπως λέγεται, ε, δηλαδή ακριβώς πριν από την αρχή της πτήσης κάθε φορά ε, θα διανεμηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις ε, τρόπος ε, ή μάλλον ένα έγγραφο το οποίο θα περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους θα γίνεται ο έλεγχος αυτός στην Ολλανδία σαν παράδειγμα η αεροπορική αστυνομία έχει την δυνατότητα να κάνει τέτοιου είδους έλεγχους έτσι ώστε να επαληθεύει τον σεβασμό της τήρησης των νομικών ρυθμίσεων που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Ε, τα επιμέρους κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα αλλά όχι την υποχρέωση να κάνουν περαιτέρω ε, μορφές ελέγχου και για άλλες ουσίες εκτός συνοπνευματοδών. Θα πρέπει όμως να ενημερώνουν την ΕΑΣΑ γι' αυτό. Και τέλος, υπάρχουν επίσης και τεχνικές ρυθμίσεις στην 15-16 του 14 σχετικά με τα συστήματα προειδοποίησης έγκαιρης, αλλά αυτά είναι τεχνικά θέματα και δεν θα ήθελα να περάσω τώρα σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Πάντως το θέμα είναι ότι οι αρχικές γερμανικές προτάσεις θα καταλήξουν τελικά στο να βοηθήσουν την βελτίωση του κλίματος ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες σας θα δώσω αμέσως τον λόγο στον Βιμ Βαντερ Κάμπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή που γίνεται σήμερα είναι πάρα πολύ χρήσιμη στα πλαίσια των ελεγκτικών διαδικασιών. Προσπαθήσουμε να δούμε το τι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΑΣΑ έχει πετύχει μέχρι τώρα. Είναι μια καλή διαδικασία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί έτσι να καταλάβει το πού πηγαίνουν τα πράγματα. Ευχαριστώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εκπροσώπους της γιατί ήταν σαφής η παρουσίαση την οποία έκαναν για τις ρυθμίσεις οι οποίες έχουν ε, αποφασιστεί μετά από το τρομερό ατύχημα που συνέβη στην ορεινή Γαλλία όπου έχασαν τη ζωή πάρα πολλοί επιβάτες μεταξύ των οποίων και πάρα πολλοί Γερμανοί μαθητές. Είναι σαφές ότι ε, θα πρέπει οι έλεγχοι που είπατε να γίνονται μόνο για τα ινοπνευματόδη ή και για άλλου είδους ουσίες και ναρκωτικά. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα το οποίο τελικά εσείς προτείνετε καλύπτει και άλλες ουσίες. Ποια είναι η άποψη της ΕΑΖΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι θα κάνουμε επίσης με αυτούς οι οποίοι υποφέρουν από κατάθλιψη. δεν είναι κάποιος ο οποίος καταναλώνει υνοπνευματόδη ε, ή ναρκωτικά, αλλά έχει κάποια προβλήματα ψυχολογικά και πολύ συχνά υποφέρει από κατάθλιψη. Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Και ένα τρίτο σημείο πρόεδρε. Είναι κάτι το οποίο άπτεται περιφερειακά του θέματος αυτού. Όταν έγινε το ατύχημα αυτό ε, υπήρξε ένα θέμα με τις πόρτες ασφαλείας του πιλωτηρίου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 Insbesondere, Βλέπω και εγώ, όπως και ο φίλος Van να μπορούμε να αποφύγουμε τέτοια φρικιαστικά σενάρια όπως η πτώση του γερμανικού αεροσκάφους, διότι εν τέλει το χρωστούμε και στην μνήμη των θυμάτων. Ιδίως θεωρώ ότι πρέπει να υποστηριχθεί η πανευρωπαϊκή υποχρέωση αεροπορικών εταιριών να δημιουργήσουν προγράμματα ψυχολογικής στήριξης πιλότων και να έχουν οι πιλότοι τη δυνατότητα να μπορούν να βρίσκουν διέξοδο από δύσκολες καταστάσεις που ενδέχεται να περάσουν στη ζωή τους ψυχολογικές ή άλλου είδους. Ως σοσιαλιστική πολιτική ομάδα ζητούμε επίσης από την ΕΑΣΑ να δημοσιεύσει το δυνατόν συντομότερο λεπτομερείς κανόνες και να εγκύψει ιδίω σε βέλτιστες πρακτικές υφιστάμενων προγραμμάτων για το θέμα αυτό. Και αν με επιτρέπετε ακόμα μια φράση για το ίδιο θέμα, θα ήθελα να επισημάνω ιδίω την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία EPPSI, που είναι Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Στήριξης Πιλότων, όπου συμμετέχουν ειδικοί ψυχίατροι, γιατροί και άλλοι και καταστρώνουν σχέδια για τέτοιε ειδικέ ε, βέλτιστες πρακτικέ. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ κύριε ΕΡΤΟΥΠ, η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πρόλαβα όλη την παρουσίαση γιατί είχα άλλη υποχρέωση, αλλά γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι και όχι μόνο για την πτώση του αεροσκάφου German Wings, αλλά και είναι πάρα πολύ αναγκαίο να γίνονται έλεγχοι της υγείας των πιλότων πρωτίστω βεβαίω από, άψη την, από την την ιατρική, των πιλότων, των κυβερνητών και συγκυβερνητών. Αλλά εδώ φαίνεται να μιλούν και για όλο το πλήρωμα του αεροσκάφους και δηλαδή ε, της αεροσυνοδούς κλπ. Πρόκειται και για θέμα ελέγχου κατανάλωσης ε, ή ε, ναρκωτικών και επειδή φαίνεται κάποια ψυχολογικά προβλήματα να έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο εκεί. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί κανείς να τον προσλάβει αυτόν ως κυβερνήτη ή ως μέλος του πληρώματο και ποιες ενδείξει υπάρχουν σχετικά με το ποιε ουσίες ενδέχεται να επιτρέπονται και ποιε όχι. Μπορούν να υπάρξουν και ψυχολογικά προβλήματα όπως και το λεγόμενο burnout. Το ερώτημα είναι μέχρι πού πηγαίνουμε και κατά πόσον επιτρέπονται οι σχετικές έρευνες για να αποκτήσει κανείς εικόνα, αν δηλαδή συμβαδίζουν με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι κάπως δύσκολη η ισορροπία. Αφενός θέλουμε οι αεροπορικές εταιρείες να γνωρίζουν τα των πιλότων, διότι δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να γίνονται πράγματα όπως αυτά με τις German Wings, όπου συμπαρέσυρε στο θάνατο που επέλεξε ο πιλότος ολόκληρο το αεροσκάφος, όλου όλους τους επιβαίνοντες του αεροσκάφους. Τώρα, αυτά ισχύουν για τους πιλότους, είπαμε, αλλά ισχύουν και για, τους, για τα μέλη του πληρώματος, τα υπόλοιπα μέσα στη μέλη του πληρώματος. Και τελευταία ερώτηση, διότι υπάρχουν και γυναίκες κυβερνήτες. Εδώ τώρα μου ήρθε αυτό. Για την ικανότητα πτήσης και κυβέρνηση του αεροσκάφους παίζει ένα ρόλο και η εγκυμοσύνη. Γνωρίζω βέβαια ότι είναι ε, σχετικά σπάνια η περίπτωση το πιδάλιο του αεροσκάφους να το κρατεί γυναίκα, αλλά νομίζω υπάρχει. Ευχαριστώ κύριε Μάσνερ. Η κυρία Κίλονεν. Ευχαριστώ αγαπητή πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρομαι ιδίως σε αυτό το βεβαίω πάρα πολύ δραματικό ε, συμβάν της ε, πτήσεως German Wings. Ε, εκτός των μέτρων που μας παρουσιάσατε, έχετε σκεφτεί ενδεχομένως αν μπορούν να ισχύσουν και άλλες διατάξεις για να συμβάλλουν στο να αποφευθούν τέτοιου είδους συμβάντα. Από την άποψη ας πούμε των τεχνικών ελέγχων. Έχετε σκεφτεί κάτι άλλο. Δηλαδή, να υπάρχει ας πούμε ε, δυνατότητα εισόδου στο κόκπιτ, στο θάλαμο διακυβερνήσεως του αεροσκάφους από αλλού και όχι μόνο από την πόρτα που προστατεύεται. Υπάρχει, έχει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκεφτεί να καλύψει ενδεχόμενα τέτοια και σε άλλες μορφές μεταφορών όπως τους ιδεοδρόμου. και αναφέρομαι κυρίως για, σε μεταφορές προσώπων, επιβατών δηλαδή. Το αεροπλάνο, το τρένο, ο σιδηρόδρομος, δηλαδή τα λεωφορεία έχουν σκεφτεί και ενδεχόμενα προληπτικά μέτρα για να αποφευθούν τέτοιες τραγωδίες στο μέλλον. Ευχαριστώ και Κίλονεν. Έχω κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις εγώ ίδια. Μιλήσατε πρώτα για ε, τεστ αλκοολεμίας που λέτε ότι δεν είναι ε, πάντοτε ακριβή. Πώς οργανώνονται αυτά. Μπαίνουν κάποια ποσοστά αλκοόλης στο αίμα, ας πούμε 0,5 γραμμάριο στο λίτρο θα είναι συνολικά δηλαδή ευρωπαϊκά αυτά ή κάθε χώρα μέλος θα θεσπίσει δικά της όρια. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Τι εννοείται ψυχολογική αξιολόγηση. Τι εννοείται πιο συγκεκριμένα. Ποιο είναι το περιεχόμενο της ε, ψυχολογικής αξιολόγησης. Είναι και θέμα ευρωπαϊκών προτύπων που να μπορεί κανείς ευλόγως να αναμένει ώστε να μπορούν να απομακρύνονται πρόσωπα τα οποία έχουν ενδεχομένω διανοητικά προβλήματα. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Και πώς θα θεσπιστούν τα πρότυπα αυτά. Θα είναι δηλαδή ευρωπαϊκά πρότυπα και πώς θα εναρμονιστούν όλα αυτά. Ο κύριος Ρικέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά όντω θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν και την ε, Τμήμα αυτό για την εργασία του. Είναι μια εργασία την οποία αναλάβατε μετά από ένα φρικτό δράμα. Ε, εγώ θέλω να μιλήσω για πρότυπα και οργάνωση. Πρώτον, ποιο αποφασίζει για τη φύση των δοκιμών. Δηλαδή, για κάθε δοκιμή, ποιο είδο ψυχο ε, δραστικής ουσίας θα ελεγχθεί για το αλκοόλ ας πούμε εντάξει αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλες ουσίες άλλες που είναι φάρμακα και άλλες που είναι ναρκωτικά Ποιος θα φτιάξει τον κατάλογο θα είναι αυτός υποχρεωτικός ή θα είναι εθελοντικό. Δηλαδή θα μπορούμε να δοκιμάσουμε ένα κομμάτι αυτού του καταλόγου. Έπειτα εξαρτάται από τη κράτη-μέλη. Εάν λοιπόν οι ε, πρακτικές είναι ασύμετρες, τι θα κάνει, θα μπορεί να τους ελέγξει, να τους παροτρύνει ή κάτι περισσότερο. Έπειτα, ποιος στα κρατημέλη ελέγχει τι γίνεται, υπάρχει αρχή και αυτή η αρχή από ποιον ελέγχεται η ίδια. Τέταρτη ερώτηση. Η Κομισιόν προτείνει μέτρα. Δηλαδή, εάν βγουν θετικές οι δοκιμές και εκεί θα εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια της κάθε εταιρεία του κράτους μέλους, είτε η Κομισιόν προτείνει μέτρα. Αν βρούμε έναν πιλότο, ας πούμε, με 2,5 γραμμάρια, ε, δεν θα το αφήσουμε να ανέβει στο αεροπλάνο. Αλλά γίνονται δοκιμές ε, στη διάρκεια πτήσεων, πριν τι πτήσει, μετά τι πτήσει, Ε, τελευταία μου ερώτηση. Θα εξασφαλιστεί ο εξαντλητικός έλεγχος, δηλαδή θα είναι τυχαίο το δείγμα ή θα ε, ρυθμιστεί έτσι ώστε το σύνολο του προσωπικού κάποια στιγμή να υπόκειται σε κάποιον έλεγχο και υπό αποδεκτές συνθήκες. Μπορεί να είμαι αλκοολικός ας πούμε και να μην με πιάσουν. Μπορεί όμως Μπορεί κάποιο τυχαία να με ελέγξει και να έχω πιει εκείνη την ημέρα, αλλά να μην είναι η συνήθειά μου αυτή ή να μην καταναλώνω αλκοόλ συνήθω. έχω Είμαστε δηλαδή σε ένα είδο ε, λίστας καλών πρακτικών και καταστάσεων όπου θα πρέπει αυτές να εφαρμοστούν ή θα διευκρινιστούν περισσότερο η φύση του προϊόντος, η φυση των προιοντων η φυση των ελέγχων και ο έλεγχος των ελέγχων. Και τέλος, για τις πτήσεις που ξεκινούν από ένα ευρωπαϊκό αεροδρόμιο, από μη ευρωπαϊκές εταιρείες θα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου για το υπτάμενο προσωπικό αυτών των εταιριών. Ευχαριστούμε κύριε Ερικέ. Ο κύριος ε, Γκόλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την ΕΑΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο έχω ένα πρόβλημα. Οι πιλότοι είναι και οδηγοί εντό εισαγωγικών. Και είναι σωστό, εάν κάποιος έχει χάσει, είναι δυνατόν κάποιος που χάνει ας πούμε το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Ε, λόγω κατάχρησης αλκοόλ ε, να διατηρεί ας πούμε το πιστοποιητικό πτήσης του, να μπορεί να ε, πιλωτάρει το αεροσκάφος. Ευχαριστώ. Ο κ. Ντελή, ευχαριστώ. Μιλούμε για τεστ. Για παράδειγμα, τεστ αίματος, αλκοολεμίας, για να ελέγξουν και ενδεχομένω και ψυχοτρόπες ουσίες στο αίμα κλπ. Μπορεί να αρνηθεί ο πιλότος ή το μέλος του πληρώματος. Γιατί σε ό,τι αφορά τα πρότυπα που προβλέπει η εργατική νομοθεσία, μπορεί κάποιος να αρνηθεί. Να αρνηθεί να υποστεί το τεστ αλκοολεμίας ή άλλης ε, ε, ενεχόμενης ουσίας. Θα υπάρχει ευκαιρία δηλαδή ο πιλότος ή το μέλος του πληρώματος να αρνηθεί να υποστεί το τεστ ή όχι και ποιες θα είναι οι συνέπειες. Μαρινέσκου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εξ όσων γνωρίζω η Κομισιόν μαζί με την ΕΑΣΑ, τέλος πάντων η Κομισιόν, συντάσσει πρόγραμμα για τους νέους κανόνες που θα απορρέουν τον βασικό κανονισμό και ελπίζω κάποια στιγμή τον Ιούνιο να δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ένωσης. Ερώτηση λοιπόν, η παράγωγη νομοθεσία που ε, αφορά το σημερινό θέμα, πότε αναμένεται. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου. Πριν να ακούσουμε τις απαντήσεις στις διάφορες και ποικίλε ερωτήσεις μας, απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να απευθύνω χαιρετισμό σε 15 σπουδαστές του Πανεπιστημίου της Λουβένης. Εσείς είστε οι φοιτητές της κοινωνιολογίας. Μην, μην τρέπεστε, σηκωθείτε. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. λοιπόν τα νεαρά αυτά πρόσωπα. Voilà, vous avez été invité par monsieur. Έχετε προσκληθεί από τον κύριο Πέλετ και καλώς ήρθατε. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε τον λόγο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ευρύ φάσμα ερωτήσεων. Πρώτα, ερώτηση για το εάν τα τεστ αναφέρονται σε αλκοολεμία ή σε ενδεχόμενη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα, γίνεται συστηματική, θα γίνονται συστηματικά τεστ αλκοολεμίας και λήψης ναρκωτικών. Δηλαδή, άμα την προσλήψει, μετά από ενδεχόμενο συμβάν, και στη βάση εύλογης υποψίας. Υπό τις συνθήκες αυτές θα γίνονται τεστ και για αλκοόλ και για ναρκωτικές ουσίες. Θα γίνονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι που δεν θα κοινοποιούνται μετά την αποκατάσταση, rehabilitation ενδεχομένως, αν δηλαδή ο πιλότος είναι κατάλληλος να κυβερνήσει το αεροσκάφος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους, το πρόγραμμα RAM ή από εθνικούς αξιωματικούς, η υποχρέωση που θεσπίζει ο κανονισμός της χώρας μέλη θα είναι να διεξάγονται τεστ αλκοολεμίας. Αυτά θα πρέπει να γίνονται λοιπόν σε όλες τις χώρες μέλη. Επιπροσθέτως, δίνεται η δυνατότητα στις χώρες μέλη, εάν επιθυμούν, να διεξάγουν και random drug testing, δηλαδή δειγματοληπτικού ελέγχου για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Χωρί να είναι υποχρεωτικό αυτό. Οι χώρε μέλη θα αποφασίσουν αν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την δραστηριότητα. Έγιναν τώρα και ορισμένε ερωτήσει για θέματα κατάθλιψης και τι μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις αυτές. Τι μπορεί να γίνει. Ε, επ' αυτού να επανέλθω σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή δεν πρόκειται για το μόνο νομοθέτημα που θα προκύψει από τις εργασίες της ε, Task Force για την ε, πτώση του αεροσκάφους German Wings. Έχουν εξετάσει επίσης και για, και άλλα όπως ε, την ιατρική εξέταση των υποψηφίων, την υποχρέωση να κοινοποιούνται ατελείς ιατρικοί έλεγχοι και άλλα σχετικά. Γίνεται μια προσπάθεια δηλαδή να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις όπως η ειδική περίπτωση του πιλότου του German Wings που ήταν καταθλιπτικός και έκρυβε την κατάστασή του από τον εργοδότη του. Το ζήτημα των ε, προγραμμάτων στήριξης είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί και θα πρέπει να χρησιμοποιείται για πιλότους οι οποίοι πάσχουν από κατάθλιψη να μπορούν να παρουσιάζονται και να ζητούν στήριξη από τους κατάλληλους ανθρώπους. Ας έρθω λίγο στις πιο εύκολες ερωτήσεις. Αν δηλαδή και άλλες εταιρείες εφόσον αυτές ξεκινούν από ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Θα χάσω την ε, άδεια πιλότου αν χάσω την άδεια οδήγηση αυτοκινήτου. Η απάντηση είναι ναι. Χωρί όμω αυτό να περιλαμβάνεται στην παρούσα γνωμοδότηση. Είναι κανόνα που υπάρχει στον κανονισμό που διέπει τα των πιστοποιητικών ικανότητας. Τώρα, η δειγματοληπτική έλεγχη θα είναι δειγματοληπτική έλεγχη στα πλαίσια του ΡΑΜ στη βάση λίστας που θα δίνει η ΕΑΣΑ. Από την άλλη μεριά, οι έλεγχοι που θα γίνονται άμα την προσλήψει και μετά από συμβάν και σε περίπτωση ευλογής υποψίας, αυτή θα είναι συστηματική. Δηλαδή θα καλύπτουν όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στις καταστάσεις αυτές. Αν θέλουν δηλαδή να ξεκινήσουν νέα σύμβαση με μια αεροπορική εταιρεία, θα ελέγχονται. Τι γίνεται εάν το τεστ αποβεί θετικό. Η πρώτη άμεση συνέπεια είναι ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν θα μπορέσει να οδηγήσει το αεροσκάφος. Δηλαδή θα πρέπει να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του ο πιλότος και θα έχει και επιπτώσεις και στην άδεια ε, χειριστού. Αυτά περιλαμβάνονται ήδη στον οικείο κανονισμό που προβλέπει και την περίπτωση κατάχρησης ουσιών. Άλλη ερώτηση αναφερόταν στο αν θα ελέγχονται πιλότοι ή και μέλη πληρώματος για τους ελέγχους για ψυχοτρόπες ουσίες, πάλι άμα τη προσλήψει μετά από συμβάν και σε εύλογη υποψία, όλα, όλα τα τεστ θα γίνονται και σε πιλότους και σε μέλη του πληρώματος καμπίνας. Ο, όποιο προσωπικό έχει σχέση με ασφάλεια του αεροσκάφους θα ελέγχεται. Ποιε θα είναι οι επιπτώσει εάν κάποιο αρνηθεί να υποστεί τον έλεγχο. τότε αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα του τεστ είναι αρνητικό με την έννοια ότι το πρόσωπο αυτό δεν επιτρέπεται να πετάξει. Και επομένως θα απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του αμέσως. Άλλη ερώτηση ήταν για το αν θα υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τα προγράμματα στήριξη, Εδώ θα παρακαλέσω τον εκπρόσωπο της ΕΑΣΑ να αναπτύξει με περισσότερα λόγια το τι ακριβώς κάνουν. Ευχαριστώ πολύ. Να σας εξηγήσω τι γίνεται με το πρόγραμμα στήριξης και πώς θα γίνεται και η αξιολόγηση. Για το πρόγραμμα στήριξης η λειτουργία του προγράμματος αυτού Βεβαίως θα λάβει υπόψη όλες τις καλές πρακτικές που ήδη ε, υπάρχουν στην Ευρώπη και χρησιμοποιούνται. Όταν αναπτύξαμε λοιπόν αυτή τη γνωμοδότηση, ε, εξετάσαμε πολύ προσεκτικά όλα τα προγράμματα στήριξης που υπάρχουν στην Ευρώπη σήμερα και διαπιστώσαμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα και μόνο πρόγραμμα για όλους. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα που λειτουργούν και αυτό θα συνεχιστεί. Ε, αυτό που έχουν κοινό είναι όλα αυτά τα προγράμματα αυτά στήριξη είναι ότι εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα. Υπάρχει όμως μια διάταξη που ορίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διερριχθεί η εμπιστευτικότητα και να δοθούν οι πληροφορίες στην αρμόδια αρχή που εκδίδει την άδεια. Όλα αυτά λοιπόν λειτουργούν αρκετά καλά σήμερα και εμείς Έχουμε, συμμετέχουμε σε αυτόν τον οργανισμό ΕΨΗ, ε, η, είναι, ε, υποστηρίζει αυτό το φόρουμ όπου ψυχολόγοι, πιλότοι και αεροπορικές εταιρείες ε, συνεργάζονται. Για την ψυχολογική αξιολόγηση είπατε ότι πρέπει να υπάρχει ίσως ένα στάνταρ ψυχολογικής αξιολόγησης στην Ευρώπη. Έχουμε δει στο σχέδιο κανονισμού ότι δεν θα πρέπει να είναι μόνο ε, μία προδιαγραφή, γιατί Υπάρχει συγκεκριμένο ψυχολογικό προφίλ για την κάθε εταιρεία για να επιλέξει έναν πιλότο. αυτό ο πιλότο θα έχει διαφορετικό περιβάλλον εργασία και ε, διαφορετικό και πίεση ανάλογα με την ε, αεροπορική εταιρεία στην οποία εργάζεται. Δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή μόνο μία ε, εκτίμηση για όλου Αυτό που είναι σημαντικό είναι να επιβλέπετε αυτό από ο ψυχολόγο που γνωρίζει την αεροπλοεία. Και αυτό έχουμε εντάξει σε αυτό το κανονισμό. Σας ευχαριστώ. Κομισιόν για όλες αυτές τις πληροφορίες και διευκρινήσεις. Ε, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Κυρία Μέσνερ, θέλετε ξανά το λόγο? Ναι, διότι με ενδιαφέρει πραγματικά τι γίνεται με τις εγγύους κυβερνήτες, δηλαδή κυβερνήτησες ας πούμε, πιλότες γυναίκες, ε, πιλότους γυναίκες. Και εσείς κύριε Βαντεν Κάμπ, ορίστε. Εγώ δεν πρόσεξα ίσως, αλλά είχα κάνει μια ερώτηση για την πόρτα του πιλοτηρίου. Κύριε Ζωακή, με θέλετε να απαντήσετε παρακαλώ. Ναι. έγκυες πιλότη, πόρτα πιλωτηρίου. Μάλιστα. Το θέμα της εγκυμοσύνης και των αγίων γυναικών δεν είναι το θέμα αυτού του κανονισμού. Υπάρχουν κανόνες στο PartMed, όπως λέγεται, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω, δεν τους γνωρίζω. Το ίδιο ισχύει και για το ερώτημά σας, το οποίο δεν ανέφερα, δεν απάντησα, το θέμα της προστασίας των δεδομένων και πάλι αυτό σχετίζεται με τους κανόνες για τα ε, κέντρα, ε, τα ιατρικά κέντρα μου ε, μόλις εγκρίθηκε. Τώρα, η πόρτα του πιλωτηρίου δεν είναι θέμα το οποίο έχουμε εδώ εξετάσει σε αυτόν τον εφαρμοστικό κανονισμό. Ωστόσο, θα ζητήσω από την ΕΑΖΑ να σας δώσει πληροφορίες για το τι συμβαίνει ε, όσον αφορά τη συνέχεια που δίνεται στην υπόθεση της πόρτας πιλωτηρίου. Σας ευχαριστώ πολύ και για την ε, πόρτα του πιλωτηρίου θα πρέπει να θυμάστε το θέμα γιατί ακριβώς μετά από το ατύχημα της German Wings η Άζα δημοσίευσε ένα φυλάδιο ε, με πληροφορίες ασφάλειας όπου συστήσαμε δύο άνθρωποι να είναι πάντοτε στο πιλωτήριο ανα πάσα στιγμή. Και αυτό οδήγησε σε πολλές ερωτήσεις, αυτή η ενδιάμεση απάντηση από τους φορείς της αεροπλογίας και έτσι κάναμε μια έρευνα στην οποία είχαν πρόσβαση όλοι οι πιλότοι, το υπτάμενο προσωπικό, όλοι όσοι συμμετέχουν ενδιαφέρονται για την αεροπλογία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περίπου 5.000 κόσμος απάντησαν στην έρευνά μας και είπαν ότι οι δύο άνθρωποι στο πιλοτούριο αυτή τη σύσταση μάλλον δεν είναι πάντοτε ο καλύτερος Τρόπο, ε, τρόπος και άρα θα πρέπει να κάνει ανάλυση κινδύνου η αεροπορική εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη διάφορα στοιχεία. Ας πούμε πόσο καλά γνωρίζει η ε, αεροπορική εταιρεία το επιτάμενο προσωπικό της, ε, ε, εάν βεβαίω έχει ε, πληθυσμό που δεν, ε, μάλλον υπαλλήλου που δεν του γνωρίζει πολύ καλά, υπάρχουν πολλέ αλλαγέ, θα ήταν ίσω καλή ιδέα να υπάρχει δεύτερη θέση και να, τόσο λεπτή και, και σημαντική θέση να μην δίνεται σε πιλότους τους οποίους δεν γνωρίζει τόσο καλά η εταιρεία. Γι' αυτό το λόγο η ΆΖΑ το καλοκαίρι του 2016 ε, δημοσίευσε άλλο φυλάδιο ασφαλείας, περί ασφαλείας μάλλον, έτσι ώστε οι πληροφορίες που έχουμε για την πόρτα του πιλωτηρίου αλλά και για τους όσους βρίσκονται εντό του πιλωτουρίου ε, αναφέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει η αεροπορική εταιρεία για το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας, λέει η Πρόεδρος. Δύο παρατηρήσεις έχω. Θα ήθελα το θέμα για τις γυναίκες πιλότους και για τις έγκυες πιλότους να μας ενημερώσετε όλους. Διότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι μέσα στις προτεραιότητές μας. Απάντηση της ΕΑΖΑ τώρα. Εγώ έχω πρόβλημα. Λέτε ότι ζητάμε από τις αεροπορικές εταιρείε να κάνουν τις μελέτες και μετά τις ε, βλέπουμε. Ναι, αλλά ο ρόλος της ΕΑΖΑ, κατά τη γνώμη μου, είναι να προβλέψει. Ίσως να μιλήσει με τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά εσείς οφείλετε να κάνετε τις μελέτες και όχι οι αεροπορικές εταιρείες, γιατί εδώ μιλάμε για την αυριανή ε, ρύθμιση. Προσέξτε το αυτό. Γιατί εγώ ως αεροπορική εταιρεία μπορώ να πω ότι δεν τρέχει τίποτα, δεν συμβαίνει τίποτα, όλα πάνε καλά, ε, αλλά εσείς θα πρέπει να ελέγξετε και άρα αυτό το θέμα είναι δική σας ευθύνη. Ίσως να έχουμε και άλλες ερωτήσεις όμως που θα σας τις στείλουμε για να συνεχίσουμε να ενημερωνόμαστε καλά πάνω σε αυτά τα θέματα. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερήσιάς μας διάταξης. Παρακαλώ, καλώς ήρθατε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Α, όχι Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Ελεκτικό Συνέδριο. Πολλοί ήρθατε μαζί. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Ζόρζε Πουφάν, που είναι ειδικό εισηγητή ε, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Έχετε 10 λεπτά. Και μετά θα ακούσουμε ερωτήσεις και σχόλια των συναδέλφων. Έχετε το λόγο λοιπόν για 10 λεπτά και βάζω και το χρονόμετρο. Καλημέρα σας, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής Μεταφορών. Οι αερομεταφορές είναι σημαντικό κομμάτι της εσωτερικής αγοράς. Ενθαρρύνει την κινητικότητα των αγαθών και των προϊόντων και των επιβατών. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των ροών στις αερομεταφορές απαιτούν την παρέμβαση για τη διαχείριση, το λεγόμενο GTA. Καταρχάς ε, κάνει τρία πράγματα, απόσταση ανάμεσα στα αεροσκάφη, εξισορρόπηση της προσφοράς ελέγχου της ε, εναέριας κυκλοφορίας, όπως επίσης και αεροναυτικές πληροφορίες στους χρήστες ε, του εναέριου χώρου. Το περιβάλλον πολλές φορές είναι μονοπολιστικό και πολυδιασπασμένο ταυτόχρονα είναι διασπασμένο με βάση τα εθνικά σύνορα, κάτι το οποίο περιορίζει την λειτουργικότητα, την ολοκλήρωση και την δυνατότητα επίτευξης οικονομιών κλίμακας. Απαιτεί επίσης για κάθε χώρα έναν παροχέα πληροφοριών, τον λεγόμενο PSNA. Όταν είναι ανύπαρκτος ο ανταγωνισμός δημιουργούνται ολιγοπόλια που επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών να δημιουργούν συνθήκες όχι υγιείς. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε καθυστερήσεις και αυξάνει το κόστος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο φυσικά καλύπτεται από τους χρήστες. Η πρωτοβουλία η ευρωπαϊκή Ουρανοί δημιουργήθηκαν για να βελτιωθούν οι επιδόσεις στη διαχείριση των εναερίων μεταφορών, μεταφέροντας κάποιες αρμοδιότητες από το διακυβερνητικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε επίσημα το 2004 και περιλαμβάνει κοινού κανόνε εφαρμόσιμού στο σύνολο της Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω και ένα πρόγραμμα τεχνολογικού εξυγχρονισμού, ε, το σχέδιο CESAR, Single European Sky ATM Research. Η πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε επίσης και με οικονομικά κίνητρα. Ο γενικός στόχος τον οποίο, ε, ε, τον οποίο έχει η πολιτική αυτή είναι η βελτίωση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των εναερίων μεταφορών. Ελήφθησαν λοιπόν νέες αποφάσεις με νέους στόχους ήδη από το 2005 και μετά, μείωση ε, κατά 50% του κόστους του GTA και μείωση 10% των αποζημιώσεων που ε, είναι απαραίτητες να δοθούν λόγω της βλάβης στο περιβάλλον στην περίοδο 2004-2020 συνολικά θα έπρεπε να φτάσουμε τα 3,8 δις ευρώ και στα πλαίσια της αναπτυξιακής φάσης των προγραμμάτων και στα πλαίσια της πλήρους εφαρμογής. περίπου δηλαδή 1,3 για την ανάπτυξη και 2,5 δις για την εφαρμογή τώρα. Εμείς πώς κάναμε τον έλεγχό μας. Καταρχάς η πρωτοβουλία του ελεγκτικού συνεδρίου έλεγξε τα συστήματα επιδόσεων, τα συστήματα τιμολόγησης, ε, τους ε, ξεχωριστούς χώρους ελέγχου και την εφαρμογή του σχεδίου ΣΕΖΑΡ και σε ποιο βαθμό όλα αυτά βελτίωσαν την αποδοτικότητα της διαχείρισης των αεραϊών μεταφορών στην Ευρώπη θα ξεκινήσει συνολικά για το πρόγραμμα ΣΕΖΑΡ ένας νέος έλεγχος το 2018. Για να ολοκληρώσουμε τον έλεγχο που κάνουμε σήμερα, ήρθαμε σε επαφή με κομβικούς οργανισμούς στον τομέα των αερομεταφορών και σε πέντε κράτη-μέλη, Ισπανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως επίσης ήρθαμε σε επαφή και με άλλους εμπλεκομένους στο λειτουργικό και βιομηχανικό κομμάτι. Τι διαπιστώσαμε. Καταρχά θεωρούμε ότι η πρωτοβουλία ενιαία Ευρωπαϊκή Ουρανού ήταν δικαιολογημένη γιατί υπήρχαν προβλήματα με τα εθνικά μονοπόλια και την πολυδιάσπαση στον βιομηχανικό κλάδο. Φαίνεται επίσης ότι τα διαφορετικά συστατικά των πολιτικών που ακολουθήσαμε έχουν σαν στόχο να διορθώσουν τα προβλήματα τα οποία είχαν σημειωθεί. Όμως οι στόχοι υψηλού επίπεδου της πολιτικής αυτής είχαν σχέση με μια περίοδο υψηλής ανάπτυξης των αερομεταφορών. Λόγω όμως της μείωσης της ζήτησης, ε, οι στόχοι αυτοί που αποφασίστηκαν το 2005 στην πρακτική δεν είναι εφαρμόσιμοι, όπως η μείωση κατά 50% του κόστους του GTA και δεν έχουν λόγο ύπαρξη σε ορισμένες περιπτώσεις όπως ο τριπλασιασμός της χωρητικότητας. Σχετικά τώρα με τις θετικές πλευρές, διαπιστώσαμε ότι το σύστημα των επιδόσεων και τιμολόγησης το οποίο δημιουργήθηκε στα πλάσια της πρωτοβουλίας βοήθησε στη δημιουργία κλίματος αποδοτικότητας και διαφάνειας στα πλαίσια των παρόχων υπηρεσιών στις εναέριες μεταφορές. Όμως υπήρξαν καθυστερήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι καθυστερήσεις αυτές είναι υψηλότερες από τα σχέδια επιδόσεων τα οποία είχαμε και δεν σταμάτησαν να αυξάνονται από το 2013 και μετά που ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο. Η μοναδιαία ή μάλλον η ενιαία μόνδα που πληρώνεται από τους χρήστες της εναέριας υπηρεσίας κάθε φορά εξαρτάται από το μέγεθος των αερομεταφορών και δεν μειώθηκε το κόστος αυτό παρά μόνο κατά 4% από το 11 μέχρι και το 16, πολύ πιο κάτω από ό,τι είχε προβλέψει η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαπιστώσαμε ότι η απουσία μιας σημαντικής μείωσης της πολυδιάσπασης που να συνοδεύεται από ποιοτικέ εξελίξεις και από λειτουργικά μπλοκ εναερίου ελέγχου δεν έχει επιληθεί ακόμα και οι μέθοδοι που ακολουθήσαμε απεδείχθησαν αναποτελεσματικές ε, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της διαχείρισης του εναερίου χώρου, της παροχής των υπηρεσιών και των τεχνικών εξοπλισμών και των δημόσιων διαγωνισμών για την κάλυψη όλων αυτών. Ε, στην ουσία έγιναν ένα αντικείμενο συνεργασίας ανάμεσα σε γειτονικέ χώρες, κάτι το οποίο δεν είναι βέβαια κακό, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο είχαμε σαν στόχο. Διαπιστώσαμε επίσης ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές έχουν δυσκολίες για να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους γιατί δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους έτσι ώστε να πετύχουν ακριβώς τους στόχους αυτούς και δεν είναι εντελώς ανεξάρτητοι από τους παρόχους των υπηρεσιών ε, ε, στον εναέριο χώρο. Σχετικά τώρα με το ΣΕΖΑΡ ε, βλέπουμε ότι έχει ενθαρρύνει τις εμπλεκόμενες πλευρές σε τεχνολογικό επίπεδο και σε αναπτυξιακή ακόμα φάση μπόρεσε να βελτιωθεί ο συντονισμός. Μια κοινή προσπάθεια όπως το ΣΕΖΑΡ δημοσιεύει σταδιακά και τακτικά λειτουργικά εγχειρίδια για την τεχνολογική και λειτουργική βελτίωση της ε, λειτουργίας ε, των υπηρεσιών αυτών. Ε, στα πλαίσια λοιπόν του πεδίου εφαρμογής και του, του πεδίου του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος αυτού τα πράγματα ε, προχώρησαν αλλά χρειάστηκε να υπάρξουν πολλές παρατάσεις. Ένα μικρό κομμάτι του σχεδίου GTA ε, έχει τελικά ολοκληρωθεί το 2016 και γι' αυτό ακριβώς η πλήρης ολοκλήρωση των προσδοκιών του ΣΕΖΑΡ έχει μετατεθεί για το 2035 και όχι το 2020 όπως είχε προβλεφθεί στο παρελθόν. Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τους στόχους υψηλού επίπεδου που έχουμε στα προγράμματα των ενιαίων ευρωπαϊκών ουρανών, ελπίζοντας ότι θα συνδυάσουν την φιλοδοξία με τις καλές επιδόσεις. Θα πρέπει πραγματικά να προσμετρηθεί και ο χρονικός παράγοντας. Θα πρέπει να αξιολογήσει επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα λειτουργικά μπλοκ εναέριας κυκλοφορίας να δούμε αν πράγματι έχουν βοηθήσει σε στρατηγικό επίπεδο. Επειδή οι εθνικές αρχές εποπτείας θα πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητες και να έχουν την δυνατότητα να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους, τα κράτη-μέλη καλούνται να καλύψουν πλήρως ε, τις ανάγκες τους τις οικονομικές και να είναι απόλυτα ανεξάρτητες πολιτικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να επανεξετάσει το σύστημα αξιολόγησης επιδόσεων και να εκλογικεύσει αν θέλετε και την διαδικασία έγκρισης των εθνικών προγραμμάτων επιδόσεων. Σχετικά τώρα με την επόμενη περίοδο αναφοράς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ελέγξει αν ορισμένοι δείκτες επιδόσεων μπορούν να τροποποιηθούν αν αυτό χρειαστεί. Σχετικά τώρα με τη βοήθεια που δίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της διαχείρισης των αερίων μεταφορών, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την συνέχιση του χρηματοδότησης αυτής με 2000, μετά το 2024, αλλά θα πρέπει να το τεκμηριώσει με τον κατάλληλο τρόπο. Θα πρέπει επίσης να δούμε και αν θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός διαχείρισης προσωρινός της κοινή πρωτοβουλία ΖΕΖΑΡ για να ενισχύσουμε ε, επίσης ε, ε, τη συμμετοχή των κρατών μελών στην κοινή προσπάθεια ΣΕΖΑΡ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καθορίσει ξεκάθαρα στάδια συμμετοχής και να καθορίσει επίσης και έναν προϋπολογισμό που να καλύπτει τα στάδια αυτά. Τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει κατά προτεραιότητα να στρέψει τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την έβρεση λύσεων που να ενθαρρύνουν την αντιμετώπιση της πολυδιάσπασης και το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αν εφαρμοστούν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, ελπίζουμε ότι θα είναι δυνατόν να έχουμε θετικά αποτελέσματα για την πρωτοβουλία ε, ε, Ευρωπαϊκή συγγνώμη, ενιαίοι ουρανοί, κάτι το οποίο θα επιτρέψει την πραγματική ενοποίηση του ευρωπαϊκού ουρανού στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ για την παρέμβασή σας που είναι πλήρης διδαγμάτων και ξεκινάμε τη συζήτηση αμέσως με τον συνάδελφο Μαρινέσκου. Κύριε Μαρινέσκου, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι σε αυτήν παρακολουθώ μάλλον αυτή την παρουσίαση, διότι παρουσιάστηκε ήδη στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Και όπως ήδη είπα, είναι πολύ καλή η έκθεση κατά τη γνώμη μου. Εντυπωσιάστηκα όταν τη διάβασα, διότι είναι πολύ σοβαρή έκθεση. Έλαβαν υπόψη όλες τις παρατηρήσεις όλων των φορέων. συμπεράσματα και συστάσεις ε, τέτοιους που θα περιμέναμε και που θα έπρεπε να γίνουν λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη και από το Κοινοβούλιο και από τους παρόχους ε, υπηρεσιών. Η Επιτροπή ε, Ελέγχου Προπολογισμού θα κάνει μια ακρόαση στις 26 Απριλίου για τον ενιαίο ουρανό. Θα καλέσουν βεβαίως και την δική μας Επιτροπή και βεβαίως και όλους όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα και με κάλεσαν στη Μαδρίτη για την συνεδρίαση της ε, ε, A6, δηλαδή του Ευρωπαϊκού, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρόχων Υπηρεσιών, για να συζητήσουν με αυτή τη μελέτη το τελικό πρόγραμμα και ελπίζω ότι μετά από αυτή τη συζήτηση και μετά και από τις ε, συζητήσεις τις πολλές που έχουμε κάνει τελευταία περίοδο θα έχουμε ίσως την ευκαιρία να ε, εισάγουμε και να παρουσιάσουμε μάλλον τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης ε, που προτείνονται από, από τα, μέρη, δηλαδή Συμβούλιο, Επιτροπή, ενδιαφερόμενους φορείς και να ανοίξουμε τις διαπραγματεύσεις για το για το πρόγραμμα, για το project αυτό που έχει παγώσει ε, όπως γνωρίζετε. Μπορούμε ίσως λοιπόν να ξανανοίξουμε το, τη συζήτηση και να βάλουμε αυτές τις συστάσεις στη νέα έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρινέσκου. Ο κύριος Έρτου θέλει το λόγο, όχι. Κυρία Μάισνερ, εσείς θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, καθώς επίσης ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον να βλέπει κανείς πώς υπολογίζεται από το ελεγκτικό συνέδριο η αποτελεσματικότητα. Πολύ ενδιαφέρον για μας. Άλλωστε, μόλις πριν λίγο ο κύριος Μαρινέσκου δήλωσε πόσο, όπως και εγώ, καιρό περιμένουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Και θεωρούμε ότι ως τώρα τα όσα έπρεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν εσφαλμένα ίσως οι στόχοι να μην ήταν σωστοί, οι στόχοι ίσως ήταν σωστοί πράγματι, αλλά οι μηχανισμοί ήταν λάθος. Λέτε ότι έχουν σημειωθεί ε, βελτιώσεις σε διάφορα πράγματα, αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Ότι ορισμένα πράγματα δεν λειτουργούν καλά, το έχουμε δει καλά, τα λεγόμενα ΦΑΠ. Είμαι Γερμανίδα. Η Γερμανία και η Γαλλία δεν χωρούν σε ένα ΦΑΠ έχουμε ξεχωριστά συστήματα και οι μεν θεωρούν τα δικά του συστήματα καλύτερα από τον δε. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο να είναι απολύτω αξιόπιστο. Γνωρίζω ότι ορισμένοι εναέροι διάδρομοι είναι και κάπως ζιγζάκ μου τα έχει εξηγήσει και ένας πιλότος από τον Μπιλμπάο μέχρι τη Φραγκφούρτη η διαδρομή είναι πραγματικά περιπετειώδης. Αυτό έχει βεβαίως και σχέση με προστατευόμενες ε, εναέριες ζώνες πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αυτά τα έχει δει το ελληνικό συνέδριο. Εγώ θα ήθελα, εκτός από το να διαπιστώσει ποια πράγματα δεν λειτουργούν, να μας πει πώς είναι δυνατόν να διορθωθούν. Είπατε ότι χρειάζεται περισσότερη δαπάνη για την έρευνα και την βελτίωση των δομών και υποδομών. Πάντως για την ώρα έχει ανασταλεί κάθε πρόοδος στον ενίο ευρωπαϊκό ουρανό λόγω της, ε, του θέματος του Γιβραλτάρ. Το καθεστώς του Γιβραλτάρ τώρα εν ώψη της Βρετανικής αποχώρησης έχει παγώσει τα πράγματα αυτά διότι είναι αβέβαιον. Τώρα, λέτε για έρευνα. Σε τι θα εστιάσει η έρευνα αυτή. Νομίζω ότι σύντομα θα χρειαστούμε νέα πρόταση. Θα ήθελα μάλιστα να ακούσω τι έχει να πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μάισνερ. Κύριε Κράμερ, εσείς. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση του θέματος. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά ευρωβουλευτή, μιλούμε για ενίο ευρωπαϊκό ουρανό, υποτίθεται ότι θα εξοικονομήσει χρήματα και θα αυξήσει την ασφάλεια. Τα θυμάμαι λοιπόν αυτά πολλά χρόνια. Ηχούν ωραία, αλλά αν κάνει κανεί μια πιο συγκεκριμένη έρευνα βλέπει ότι αυτά δεν γίνονται. Όπως είπε και η κυρία Μάισνερ, α, μας λέμε και εμείς οι Γερμανοί, Α, όχι. Εκεί οι εθνικοί εγωισμοί είναι ισχυρότεροι και από τις ενδεχόμενες εξοικονομήσεις. Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα. Τα εξετάσατε εσείς αυτά ως ελεγκτικό συνέδριο. Θα ήθελα να μου πείτε με συγκεκριμένα παραδείγματα πού έγιναν εξοικονομήσεις συγκεκριμένα πόρων. Υπάρχει κάποια χώρα η οποία μπόρεσε να διασυνδεθεί με άλλες με τέτοιο τρόπο μέσω του ευρωπαϊκού ουρανού ώστε να μπορέσει να εξοικονομήσει προσωπικό ή υποδομές. Θα ήθελα επίσης να μάθω εγώ βλέπω δηλαδή τους εθνικούς εγωισμούς να είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Έχετε κάποια θετικά παραδείγματα όπου χώρες μέλη συνεργάστηκαν και μπορείτε να μας πείτε ναι έγινε και τα πράγματα πήγαν ως εξής. Μπορείτε να μας πείτε και με ονόματα ποιοι μπλοκάρουν παρόλο που υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά αυτά τα πράγματα είναι εγκεκριμένα και έχουν εγκριθεί και με την υπογραφή των χωρών μελών, οι οποίε ξαφνικά τα έχουν ξεχάσει, διότι πάντα ψάχνουν και βρίσκουν ένα παραθυράκι, μια διέξοδο, για να μην το αφήσουν να λειτουργήσει το σύστημα. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Κύριε Ποφάνα, θα στρέφομαι σε εσά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μπορώ να σας πω ότι για να συντάξουμε αυτή την έκθεση δουλέψαμε πολλού. Είναι πολύ. Δεν ήταν εύκολη η υπόθεση. Το 2017 τον Ιανουάριο επισκεφθήκαμε ε, παρόμοιες θεσμούς ε, το ελεκτικό συνέδριο των ΙΠΑ. General Accounting Office και μα κάλεσαν εκεί για να ανταλλάξουμε εμπειρίε, γιατί οι Αμερικανοί έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται LegGen και είναι παρόμοιο με το Caesar και το συζητήσαμε εκεί, αλλά και στο Υπουργείο Μεταφορών, αλλά και με την Αμερικανική Αρχή Αεροπλοίες, με τους ε, υπαλλήλους εκεί, ώστε να κάνουμε μια μικρή σύγκριση ανάμεσα στη δική μας πρόοδο και το τι έχουν κάνει στις ΗΠΑ. Με την ευκαιρία αυτή, με την επίσκεψη αυτή, Μας είπαν λοιπόν πως ήταν καλύτερο για μας όταν θα συνεχίζαμε την έκθεση το 2018 να επισκεφτούμε τον Καναδά. Γιατί τον Καναδά, γιατί η Καναδοί είναι καλύτερη στην ε, διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας. Το αναγνώρισαν αυτό οι Αμερικανοί και ε, ευτυχώς γιατί εκεί μπορούμε να βρούμε, να ε, βρούμε έναν κύριο που είναι ο Γενικός Διευθυντής της Air Canada. Ελπίζουμε ότι θα κάνουμε αυτή την επίσκεψη ε, μέσα στους επόμενους μήνες για να έχουμε μια επιπλέον εμπειρία όσον αφορά τον ελληνικό ευρωπαϊκό ουρανό. Για τις μετακινήσεις, στους διαδρόμους των αεροπλάνων, να σας πω ότι η ομάδα μου μετέβη στην Σουηδία και όταν επέστρεφε στο Λουξεμβούργο, κανονικά η ε, διαδρομή πρέπει να διασχίσει την Γερμανία. Αλλά επειδή το κόστος στη Γερμανία για μία ώρα για να πληρωθούν οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας είναι ψηλό, είναι καλύτερο να περάσουν από την Τσεχία. Πρέπει ωστόσο να πληρώσουν το καύσιμο από την άλλη πλευρά και διαρκεί κάπως περισσότερο, αλλά βγαίνει φθηνότερα. Οι πιλότοι και οι αεροπορικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να επαληθεύουν ποιες είναι οι φθηνότερες διαδρομές. και δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι χώρες που έχουν κάνει μια διαφοροποιημένη πολιτική και ποιες είναι αντίθετες. Είναι δύσκολο να το κάνουμε αυτό, γιατί σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα υπάρχουν τώρα 28 σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα οι αρχές, ας πούμε στη Ρουμανία ε, λέγεται Ρωμάτζα η αρχή και κάθε αρχή εθνική ασκεί τη δική της πολιτική. Είναι δύσκολο να έχουμε μια γενική και συνεχτική εικόνα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Και θα συνεχίσουμε τώρα στην ημερήσια μας διάταξη. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, σας ευχαριστούμε που μας κάνετε αυτή την εισήγηση. Βεβαίως είναι η εκθεσή σας ένα θέμα, όπως το είπατε κύριε Μαρινέσκου, που θα μας απασχολήσει γιατί είναι πολύ σημαντική δουλειά και σοβαρή δουλειά, αλλά και τα αιτήματα που υποβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαβιβαστούν. Δεν τα συζητήσαμε αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ρόλος μας ως νομοθέτη είναι να τα διαβιβάζουμε. Ε, πάση σε περιπτώσει είστε ευπρόσδεκτοι εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάσσουμε απόψεις τακτικά και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την παρουσίασή του. Θα συνεχίσουμε τώρα τις εργασίες μας με το επόμενο θέμα που είναι ο χειρισμός των ε, οχημάτων με κινητήρα μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου. Κύριε Αρτούκ, εσείς είστε ο εισηγητής και έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πριν εισέλθω στο θέμα θα ήθελα να μάθω εάν είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Είναι παρούσα εκπρόσωπος ή παρόν εκπρόσωπος για ποια γενική διεύθυνση. Ναι, είναι παρούσα η γενική διεύθυνση MOVE. Α, δεν έχει έρθει ακόμη ο εκπρόσωπος. Λέτε να περιμένω ή να προχωρήσω αμέσως. Όχι, αρχίστε, αρχίστε κύριε Τούγκ με την παρουσίαση της εκθέσεώς σας. Καλά, ναι, τέλος πάντων, λέει ο κ. Σερτούγκ. Κοιτάξτε, ας αρχίσω εκφράζοντας πρώτα τις ευχαριστίες μου σε όλες και όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής Μεταφορών, διότι φάνηκε ότι η επικοδομητική συζήτηση που διεξήχθη κατά την παρουσίαση της εκθέσεως απηχείται και στις τροπολογίες όπου έγιναν κυρίως ουσιαστικές συμπληρώσεις που κάνουν το περιεχόμενο της εκθέσεως πιο σαφές. Έχω ορισμένες σχετικές παρατηρήσεις που αναφέρονται και στην ουσία. Αφενός νομίζω ότι το πιο σημαντικό για όλες και όλους τους συναδέλφους είναι το θέμα της τράπεζας δεδομένων. Άλλωστε, αυτό έδειξε και η συζήτησή μας, ότι δηλαδή δεν επιθυμούν καθε αυτήν τράπεζα δεδομένων και αναζητούν άλλες λύσεις. Εγώ συμφωνώ. Η λύση δηλαδή θα πρέπει να λάβει τη μορφή ώστε οι τράπεζες δεδομένων εφόσον υπάρχουν στο επίπεδο κρατών μελών να διασυνδεθούν, να δικτυωθούν, να θεσπίσουμε κοινά πρότυπα για να είναι δυνατόν να γίνεται ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τραπεζών αυτών. Εάν δεν επιθυμούμε λοιπόν Ευρωπαϊκή Τράπεζα Δεδομένων και εφόσον αυτό το αποφασίσουμε μπορούμε να προχωρήσουμε ταχύτερα διότι προσωπικά και νομίζω και άλλοι εδώ ενδιαφέρομαι να μπορέσει να μπει ένα τέλος στις απάτες των ταχογράφων. Για τις τεχνικές λύσεις τώρα, ορισμένοι συνάδελφοί μου, αλλά και εγώ προσωπικά, προτείνουμε τα κριτήρια, μάλλον ακριβή καθορισμό των κριτηρίων για την παραποίηση των δεδομένων των ταχογράφων. Το άλλο σύνολο διατάξεων, blockchain λέγεται, Λέει, η τεχνολογία να υπαχθεί πρώτα σε μια ανάλυση κόστους ωφέλους. Συμφωνώ, διότι χρειάζεται μια επιστημονική, οικονομολογική βάση για να αποδείξει την αξία της ρύθμισης αυτής. Και το επόμενο ε, πλαίσιο θεμάτων είναι το χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να τηρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και πριν λάβω τον λόγο ρώτησα εάν είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών συμφωνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δράσει ταχύτατα και γι' αυτό θα ορίσουμε προθεσμία 12 μηνών. Και μιας και έχουμε φτάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιτρέψτε μου να πω μια φράση ακόμα, που παρακαλώ να μην παρανοηθεί από τις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής, που μέχρι τώρα φάνηκαν πολύ συνεργάσιμες και ανοιχτές απέναντι στη δική μας εργασία. Τα τελευταία, μάλλον τους τελευταίους μήνες και εβδομάδες, ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω και παρακαλώ να σημειωθεί στα πρακτικά ότι τουλάχιστον τέσσερις γενικές διευθύνσεις παραπέμπουν το θέμα ημέν στις δε. Το λέω αυτό γιατί δεν μπορώ να το πω και διαφορετικά. Ασφαλώς συχνά έχουμε συνομιλήτρια μας στην Γενική Διεύθυνση MOVE, με την οποία έχουμε πολύ θετικές επαφές. Όμως, για το συγκεκριμένο θέμα έχουμε επαφές και με τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Just, και με την Connect, καθώς και την Growth. Αυτό δεν μας διευκολύνει. Εάν δηλαδή το θέμα μας, όταν μάλλον θέλουμε να θέσουμε το θέμα μας, να μας λένε «Α, δεν είναι αρμόδια η δική μας Γενική Διεύθυνση, πηγαίνετε στην επόμενη» προσπαθούμε με πολύ κόπο να μάθουμε ποιο είναι τέλο πάντων ο αρμόδιο στη συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση, μόνο και μόνο για να ξανακούσουμε ότι ούτε αυτή είναι η αρμόδια Γενική Διεύθυνση και α πάμε να απευθυνθούμε αλλού. Και όταν τελικώ καταλήξαμε ποια Γενική Διεύθυνση θα πρέπει κανονικά να είναι αρμόδια, σύμφωνα με τα όσα μα είχαν πει οι προηγούμενε. δεν λαμβάνουμε απάντηση επί ένα μήνα. Τα λέω αυτά με καθαρά λόγια, διότι δυσχεραίνει πολύ το έργο μας και τη συνεργασία μεταξύ, ευρωπαϊκών θεσμών και είναι απαράδεκτο ως συνομοθέτες να αντιμετωπιζόμαστε με τέτοια μεταχείριση. Ελπίζω λοιπόν ότι από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση κάποιος είναι σήμερα παρόν. DG Just και να μπορέσει να δηλώσει εάν όντως η DG Just είναι αρμόδια για να καταθέσει νομοθετική πρόταση εδώ, παροιμήν, στην Επιτροπή Μεταφορών. Αν δεν συμβαίνει αυτό θα θέλω να μου δηλώσει καθαρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιο είναι υπεύθυνο συγκεκριμένα για να μα δώσει κάποια απάντηση. Ούτως ή άλλω υποχρεούται η αλλω υποχρεουται η Επιτροπή να μα δώσει απάντηση μέσα σε μια συγκεκριμένη προθεσμία. Αυτά τα λένε και οι συνθήκε. Ωστόσο σίγουρα θα είναι σκόπιμο και χρήσιμο να ακούσουν και οι άλλοι συνάδελφοί μου ποιος είναι ο παραλήπτης της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας την οποία έχουμε συντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ζόρς. Μόλις έφτασες, αμέσως ε, σε βάλαμε στο στόχαστρο. <laughs> Ε, ευχαριστώ λοιπόν, λέει ο κύριος Μπαχ, ε, Ευχαριστώ τον εισηγητή. Δεν πρόλαβα να ακούσω τι δήλωσε, αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Πάντως, γενικά, οι τροπολογίες κατευθύνονται λίγο πολύ όλες στην ίδια κατεύθυνση και αποσκοπούν επιτέλους την ανάλυση συγκεκριμένη δράση κατά της παραποίησης των ε, ενδείξεων των ταχογράφων στα αυτοκίνητα. Έχει έρθει πια η ώρα να ρυθμίσουμε το θέμα αυτό υπέρ των καταναλωτών. Και αυτό είναι σημαντικό να το πει η έκθεση και να το υποστηρίξει. Είναι σημαντικό οι αγοραστές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων να έχουν πρόσβαση στα συγκεκριμένα δεδομένα. Εάν ερμηνεύω σωστά τις τροπολογίες, βλέπω ότι η πλειονότητά του στάσεται υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού πλαισίου, ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα, αλλά και μηχανισμοί συλλογής των δεδομένων. Εγώ είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτή την προσέγγιση. Ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί ακόμα είναι μέσα σε, ποιο, σε ποια χρονική περίοδο θα πρέπει να τα συντάξει αυτά, τις προτάσεις αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για αυτό το χρονικό πλαίσιο θα χρειαστεί ακόμη να συζητήσουμε. Και δύο λόγια τώρα για τις τεχνικές επιθεωρήσεις, PTI. Θεωρώ ότι μια μείωση της ισχύω της πρώτης τεχνικής επιθεώρησης ε, δεν λύνει κανένα πρόβλημα, γιατί υπάρχει, πάντα θα υπάρχει μια απόσταση. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε συντήρηση του οχήματος να σημειώνονται τα σχετικά δεδομένα, δηλαδή τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Τώρα για το λεγόμενο blockchain και άλλες τεχνικές δυνατότητες καταγραφής του αριθμού των χιλιόμετρων. Πάλι εκεί νομίζω ότι οι τροπολογίες κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Θα πρέπει πάντω να δοκιμαστούν αυτές οι τεχνολογικές λύσεις. Εάν στο μέλλον προκύψει μια τεχνολογικά ασφαλής μέθοδος για την διαβίβαση των δεδομένων, να την χρησιμοποιήσουμε. Μέχρι τότε όμως ας αναζητήσουμε ρεαλιστικές λύσεις. Ευχαριστώ, συνεργάζομαι με τον εισηγητή και με τους άλλους συναδέλφους και θεωρώ ότι πάντως πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στη σύνταξη ενός στέρεου κειμένου. Ευχαριστώ. Μάκερ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον, τους συναδέλφους ε, σκιώδης εισηγητές και όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στην εξέταση αυτού του θέματος. Φαίνεται πως υπάρχει συνένεση στο κοινοβούλιο μας όσον αφορά τον επίγοντα χαρακτήρα αυτού του προγράμματος, δηλαδή ε, την... Ε, την παραποίηση δεδομένων. Εγώ ε, υπέβαλα κάποιες ε, τροπολογίες μαζί με τον με τον συνάδελφο Βοσέλτε. Για μας ε, πολύ σημαντικό είναι να βρεθεί λύση σύντομα, μια αποτελεσματική λύση και μάλιστα σύντομα. Και όσον αφορά τις, το κόστος Μπορεί το blockchain να είναι κάποια λύση. Πάντως για την ώρα φαίνεται να είναι στο μέλλον όλα αυτά. Αν θέλουμε πραγματικά να εξυπηρετήσουμε τον Ευρωπαίο ε, ε, πολίτη και καταναλωτή, θα πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένη και απτή ε, απάντηση. Και η απάντηση μου φαίνεται προφανής. Υπάρχουν ήδη συστήματα στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Υπάρχει το CarPass στο Βέλγιο και αντίστοιχα συστήματα και στην Ολλανδία που μπορούν να καταγράφουν συστηματικά με αξιόπιστο τρόπο τα χιλιόμετρα και μάλιστα σε συγκεκριμένη συχνότητα. Θα μπορούσε ίσως αυτό τα τα στοιχεία να αποθηκεύονται στις εθνικές βάσεις δεδομένων. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια υπάρχοντων ε, μέσων και ε, μετρητών, θα μπορούσαμε να καταγράφουμε αυτά τα χιλιόμετρα, θα μπορούσε οποιοδήποτε, ε, διάφοροι δηλαδή οργανισμοί, διοίκηση, να ελέγχουν αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι κάτι το εξαιρετικά δαπηρό, είναι μια απλή χρήση των όσων ήδη υπάρχουν. Είναι ένα θέμα λοιπόν για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δείξει την προστιθέμενη της αξία στα, κατευθείαν στους πολίτες, γιατί αυτό εδώ το ζήτημα επηρεάζει τα καθημερινά τους προβλήματα. Και όπως είπα, χωρίς να δημιουργηθούν ε, ε, νέοι κανόνες, υπερβολικοί νόμοι κτλ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αγγίζει ένα σωρό κόσμο και ελπίζω πραγματικά πως η Κομισιόν θα λάβει υπόψη αυτό μας το μήνυμα και ότι θα μας ακολουθήσει ώστε να δώσουμε αυτό το ε, ισχυρό μήνυμα προς τους πολίτες μας. Μαζί με τους συναδέλφους λοιπόν θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ντέμις Μέκερα. Ο κύριο Ρικέ, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Ισμαήλ για αυτή την έκθεση που είναι εξαιρετική. Πάντοτε έχει την τύχη να δουλεύει σε εξαιρετικές εκθέσεις και δεν έχουμε να πούμε και πολλά λόγια. Όταν είναι καλή εκθέση όμω δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Οι κακέ εκθέσεις μα δίνουν για πιο πολύ ώρα τον λόγο. Πρώτη μου παρατήρηση. Κανένα δεν αμφιβάλλει ότι η παραποίηση των ε, μετρητών ε, ε, χιλιόμετρων είναι απάτη και έπειτα έχει και συνέπειες επιπλέον ασφάλειας. Τα κράτη-μέλη όμως δεν ενδιαφέρονται καθόλου και απόδειξη γι' αυτό είναι ότι καμιά δεκαριά κράτη-μέλη δεν τιμωρούν καν αυτό το γεγονός και εκτός από δύο χώρες οι υπόλοιπες δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Και αυτό γιατί, γιατί δεν αφορά αυτό την τσέπη των κρατών μελών, αλλά την τσέπη των πολιτών. Από τη στιγμή που κλέβονται μεταξύ τους οι πολίτες, οκ, από τη στιγμή που δεν κλέβουν την εφορία. Απίστευτο είναι ένα, μια τέτοια πάτη που είναι ε, πολύ σημαντική, αλλά και επικίνδυνη, να μην ενδιαφέρει κανέναν από τα κρατημέλη και να έχει χρειαστεί αρκετό χρόνος για να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό η Ένωση. Γι' αυτό τον λόγο μάλιστα προτείναμε όπως και σε πιο στεναρά ε, ε, μέτρα, πιο ισχυρά μέτρα, γιατί άμα περιμένουμε την καλή θέληση των κρατών μελών, ε, ζήσε μάη μου. Για το, για το blockchain έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Ε, η επιφύλαξή μου είναι ότι είναι ότι καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια και ότι αν αρχίσουμε να φτιάχνουμε μάλλον να ε, προχωρούμε σε αυτή την κατεύθυνση, τη τεχνολογία του blockchain, περνάμε σε μια ιδιαίτερη κατάσταση γιατί μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για ένα σωρό άλλε βάσει δεδομένων. Και αυτό θα πρέπει να το μελετήσουμε από ενεργειακή και οικολογική πλευρά. Και κάτι άλλο που με ενοχλεί πολύ είναι ότι από τη στιγμή που μπαίνουν τα στοιχεία στο blockchain δεν μπορεί να κάνεις πίσω και αν υπάρξει λάθος από κάποιο χειριστή αυτό θα είναι πρόβλημα, γιατί οι ε, υπάλληλοι που το χειρίζονται δεν είναι τίποτα επίσημοι ή κυβερνητικοί υπάλληλοι, είναι οι ε, συντηρητές των αυτοκινήτων, ε, στα γκαράζ κτλ. Μπορεί να θεωρηθεί λοιπόν επίσημη βάση δεδομένων το blockchain. Εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις. Νομίζω πως ε, δεν θα έχουμε ωστόσο ε, δυσκολίες να φτάσουμε σε μεγάλη συνένεση, να είμαστε όμως αρκετά αυστηροί ώστε να πιέσουμε την, κράτη, την Κομισιόν να επιβάλλει στα κράτη-μέλη ε, αυτόν τον έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρικέ. Ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ βεβαίως τον εισηγητή. Και διαρωτώ κοιτάξτε, μια έκθεση όπου δεν χρειάζεται να γκρινιάξω. Μήπως κάτι δεν πάει καλά, είτε εσύ είτε εγώ. Και εδώ μάλιστα στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει πραγματική συνένεση. Λέμε ότι καταδικάζουμε την απάτη, καταδικάζουμε τις χώρες μέλη, καταδικάζουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι έχουμε κάνει ερώτηση ως Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρεται σαν να έχει άπειρο χρόνο στη διάθεσή της. Χρειάστηκε λοιπόν να αναλάβουμε εμείς να κάνουμε έκθεση πρωτοβουλίας, διότι πρόκειται για περιπτώσεις απατών που πρέπει να απαγορευτούν. Και βεβαίω είναι και θέμα ασφαλεία, όπω είπε και ο κύριο Ρικέρ. Εάν αγοράσω ένα αυτοκίνητο που έχει πάνω από 100.000 χιλιόμετρα και εγώ τελώ στην πεποίθηση ότι έχει μόνο 25.000, κινδυνεύω. Ενώ δαπανούμε αλλού πολλά χρήματα, εδώ δεν κάνουμε απολύτω τίποτα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και ούτε χρειάζεται καν να εφεύρουμε εκ νέου τον τροχό. Βέλγιο και Ολλανδία δείχνουν σε όλη την Ευρώπη και αν θέλετε και στον κόσμο πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί. Και εμείς δεν είμαστε καν σε θέση εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πείσουμε τις άλλες χωρισμένοι να αντιγράψουν το σύστημα αυτό, να το μιμηθούν, να το κοπιάρουν, δεν επιτρέπεται να μπαίνουν μπροστά οι εθνικοί εγωισμοί. Βεβαίω και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασία προσωπικών δεδομένων. Αλλά δεν είναι πρόβλημα αυτό. Δεν θέλουμε να μάθουμε πού πήγε ο κάθε οδηγό και πότε. Όταν το αυτοκίνητο πηγαίνει στο συνεργείο, όπω γίνεται στο Βέλγιο και στην Ολλανδία, ή στο τεχνικό έλεγχο, σημειώνει το αριθμό των χιλιόμετρων. Τελείωσε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι εξαγωγέ εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτό. Και αυτό πρέπει να ελέγχεται. Διότι Εάν δεν συμβεί αυτό, τότε βεβαίως γίνεται αρνητική η εικόνα τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Οι Αφρικανοί θα πούν, α, μάλιστα, δεν επιτρέπεται Ευρωπαίοι να εξαπατούν Ευρωπαίου, αλλά επιτρέπεται να εξαπατούν του Αφρικανούς. Και τότε κάνουμε μεγάλη ζημιά στην αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωση. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Σα ευχαριστώ για την θαυμάσια εκθεσή σου Ισμαήλ. Δεν περίμενα να τα καταφέρει ο μεγάλος συνασπισμός ο ευρύ συνασπισμό στη Γερμανία. Τόσο γρήγορα, τόσο καλά, αλλά μπράβο. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Ο κύριο Κόχ. Αγαπητέ Ισμαήλ, ευχαριστήσεις και από μένα. Τρία σχόλια. Στις τροπολογίες μου αναφέρομαι πρώτα στις επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια των απατών γύρω από τους ταχογράφους. Διότι η παραποίηση υποσκάπτει την ασφάλεια χρήση του οχήματο. Δεύτερο, χρειάζεται ένα χρονικό πλαίσιο. Γι' αυτό προτείνω μέχρι τέλους του 2019 να δημιουργηθεί νομικό πλαίσιο για να δυσχεραθεί, να γίνει πιο δαπανηρή η απάτη των ταχογράφων. Εσύ προτείνεις 12 μήνες, νομίζω ότι πραγματικά βρισκόμαστε πολύ κοντά. Τρίτο, είναι σωστό να προταθούν νέες τεχνολογίες για το μέλλον που να αποκλείουν την παραποίηση η αλλίωση των δεδομένων ή να την δυσχεραίνουν σημαντικά, αλλά νομίζω ότι όλες οι χώρες μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν πρώτα το θαυμάσιο πρότυπο Βελγίου και κάτω χωρών που τα ακούσαμε. Να υπάρχουν μητρώα όπου θα καταγράφεται ο αριθμός των διανυθέτων χιλιόμετρων σε κάθε είσοδο του οχήματο στο συνεργείο και όχι μόνο στην πρώτη ε, είσοδο. Θα χαρώ πολύ να μπορέσεις να δεχτείς κάποιες από τις δικές μου τροπολογίες και να τις συντάξεις στις συμβιβαστικέ σου. Van Miltenberg. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή για μια εξαιρετική πρόταση. Έχουν κατατεθεί αρκετές τροπολογίες και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον το οποίο προκαλεί. Είναι λοιπόν μια σημαντική στιγμή για την εμπιστοσύνη την οποία πρέπει να δείχνει ο πολίτης και για την δυνατότητα που έχουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουμε να δράσουμε θετικά αναφερόμαστε στα θετικά παραδείγματα των κάτω χωρών και του Βελγίου και θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην αποφεύγει να πάρει απόφαση και να καταλήξει το ταχύτερο δυνατόν σε μία νομοθετική πρόταση. Όπως είπε ο κύριος Ρικέ, καταθέσαμε τροπολογίες έτσι ώστε μέσα σε ένα χρόνο να υπάρξει επιτέλους μία νομοθετική πρόταση. Θέλουμε να υπάρξει σωστό συντονισμός ανάμεσα στις γενικές διευθύνσεις γιατί το θέμα αυτό είναι κάτι το οποίο θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και έχουμε και το κέντρο έρευνας και τεκμηρίωσης ε, που θα μπορέσει να βρει ακριβώς που υπάρχουν κενά και πώς μπορεί να καλυφθούν. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Βαν Μίλτενμπουργκ. Α, ο Βάντερ Κάμπφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τις ανησυχίες τις οποίες εξέφρασε ο Ισμαήλ Ερτούγκ το κοινοβούλιο εδώ στην ουσία το παραπέμπωνε από τη μία γενική διεύθυνση στην άλλη και η Επιτροπή δεν έχει καμία διάθεση να πάρει απόφαση. Τέσσερις γενικές διευθύνσεις μεταξύ τους δεν μπορούν να συμφωνήσουν, η κατάσταση λοιπόν είναι απαράδεκτη και απευθύνω έκκληση στην DG Move να ξεκαθαρίσει επιτέλους τις αρμοδιότητες της κάθε ε, διεύθυνσης εμείς σαν συντονιστές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ήδη στείλαμε μια επιστολή απαιτώντας να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, να ρωτήσω τον εισηγητή εδώ κάτι. Ε, ποιοι είναι οι στόχοι σας βράχη πρόθεσμα και ποιοι είναι οι στόχοι σας μακροπρόθεσμα. Νομίζω ότι έχει σημασία ε, να δούμε αν θα ε, επιλέξουμε ας πούμε την ε, βελγική πρόταση ή μήπως θα έπρεπε να επιλέξουμε το blockchain, το οποίο βέβαια είναι πιο απαιτητικό. Αλλά δεν θα πρέπει να αναμειγνύουμε τις βαχυπρόθεσμες προτάσεις με τις μακροπρόθεσμες και αν κατάλαβα καλά την έκθεση του κυρίου Ερτούγ, αυτοί οι οποίοι θα φυγούν περισσότερο είναι οι ασθενέστεροι οικονομικά και ακόμα και η μεσαία τάξη επίσης θα φυγεί. Ε, αναφερόμαστε πάρα πολύ και στη Γερμανία στα πλαίσια του μεγάλου συντονισμού στην μεσαία τάξη η οποία έχει ε, να πολλά προβλήματα και στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Βιμ Βαντερκάμπ. Ως πρόεδρος θα ήθελα να πω στον συνάδελφο Έρτουγκ ότι πράγματι θα πρέπει να τον συγχαρώ γιατί πράγματι το έγγραφο αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προκαλέσει επιτέλους την προσοχή μας. Δεν είναι μόνο θέμα δικαιώματος των καταναλωτών, αλλά είναι θέμα κυρίως εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Εμείς δεν έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις να δώσουμε, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει συγκεκριμένες απαντήσεις να μας δώσει. Υπενθυμίζει ο κύριος Σέρτουγκ ότι στο Βέλγιο και στις κάτω χώρες είναι λειτουργικά τα συστήματα. Ε, γιατί να μην εναρμονίσουμε λοιπόν τα συστήματα αυτά και στην υπόλοιπη Ευρώπη και να τα εφαρμόσουμε. Υπάρχει απάτη στην Ευρώπη ως προς αυτό. Είναι σαφές και θα πρέπει να την λάβουμε υπόψη μας. Ζητώ λοιπόν από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης MOVE, να μας δώσει πλέον συγκεκρισμένες απαντήσεις και να μας πει τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εξακολουθεί να περνάει ο καιρός υπάρχει ένα, μια προσπάθεια ξεφορτώματος του προβλήματος από τη μία γενική διεύθυνση στην άλλη και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου τα δικαιώματα των καταναλωτών θίγονται και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και αυτή μικραίνει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε το θέμα αυτό είναι αρκετά περίπλοκο γιατί καλύπτει πράγματι διαφορετικούς τομείς. Εμείς κάνουμε σε εσωτερικό επίπεδο ό,τι μπορούμε για να δούμε τι μπορούμε πραγματικά να προτείνουμε. Εγώ είμαι υπεύθυνη για θέματα οδικής ασφάλειας. Θα ήθελα να πω ότι εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει, και μετά θα πρέπει και η Γενική Διεύθυνση για την Ανάπτυξη να εκφράσει τις δικές της απόψεις σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται ε, για την έγκριση τύπου και έχουμε και επαφή με συναδέλφους με την Γενική Διεύθυνση Δικαίου έτσι ώστε να ε, προχωρήσουμε στο νομικό πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή. Σχετικά τώρα με τις ε, τεχνικές προδιαγραφές, αυτό το οποίο ήδη είπα την προηγούμενη φορά είναι ότι συμφωνούμε με τις απόψεις σας και εμείς ε, θέλουμε να προχωρήσουμε στην δημιουργία ενός συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών ηλεκτρονικών. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα καλύψει πολλά προβλήματα και στον τομέα των απατών στους χιλιομετρητές. Υπάρχει κάτι εδώ το οποίο θα πρέπει να διευκρινίσουμε σχετικά με τη διατύπωση της ε, τροπολογίας 14. Δεν υπάρχει άμεση σύνδεσμο, άμεσος σύνδεσμος ανάμεσα στα τεχνικά χαρακτηριστικά από τη μία ε, και τον χιλιομετρητή από την άλλη. Όταν περάσει τεχνικό έλεγχο, ένα όχημα θεωρείται ασφαλές για να κυκλοφορήσει ανεξαρτήτως αυτού που γράφει ε, στον, οδομετρη, στον ε, χιλιομετρητή. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τη σημασία της τροπολογίας 46 και να διευκρινίσω εδώ ότι υπάρχει μια προθεσμία την οποία έχουν θέσει οι δύο συνομοθέτες σχετικά με την οδηγία για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων. Το ίδιο σχόλιο θα κάνουμε και για την τροπολογία 86 είναι κάτι το οποίο καλύπτεται από το άρθρο 86 συνολικά της προηγούμενης οδηγίας σας. Σε αυτή τη φάση δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Εξετάσαμε προσεκτικά την έκθεση και τις τροπολογίες τις οποίες έχουμε καταθέσει. Γνωρίζουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, επαναλαμβάνουμε αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη συνάντηση. Έχουμε κάνει το πρώτο βήμα θα ήθελα να κάνω τρεις συγκεκριμένες, μάλλον γενικού τύπου δηλώσεις. Καταρχάς θα πρέπει να βρούμε τη νομική βάση. Όπως πολύ σωστά είπατε εδώ στην πρότασή σας ε, υπάρχει απέτηση να γίνει κάτι τέτοιο για λόγους ασφαλείας. Δεύτερον, ε, βασικός στόχος της ε, νομοθετικής μας ρύθμισης σχετικά με την ε, έγκριση τύπου είναι η λεγόμενη ουδετερότητα της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας. Και αυτό καλύπτει και θέματα ασφαλείας σχετικά με τους χιλιομετρητές. Βέβαια θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι για να το πετύχουμε αυτό με τον σωστό τρόπο, απαιτούνται μελέτες και απαιτείται υιοθέτηση σωστών μορφών ελέγχου. Ευχαριστώ πολύ. Την Επιτροπή και τώρα θα πρέπει να σας πω ότι δεν μ' αρέσουν καθόλου οι απαντήσεις σας. Δεν με ικανοποιούν καθόλου. Διότι το να μου λέτε προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και μετά να ακούμε διάφορες γενικές σπουδαίες δηλώσεις επί της αρχής δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν έχουμε να κάνουμε ένα φαινόμενο που παίρνει σημαντικές διαστάσεις σε ορισμένα κράτη. Ελπίζω λοιπόν ότι η έκθεση του συναδέλφου Ερδούκ που θυμίζω θα εγκριθεί στις 25 ε, Απριλίου θα σας αναγκάσει να ξαναεξτάσετε την κατάσταση και να μας υποβάλλετε σύντομα στους νομοθέτες ένα πλαίσιο για να προχωρήσουμε. Σας το λέω έτσι κάπως άμεσα, αλλά νομίζω πως σε αυτή τη θητεία μπορούμε ακόμα να μελετήσουμε κείμενα που και να δώσουμε απαντήσεις συγκεκριμένες. Και να μην χασομεράμε εδώ, εφού, εδώ και χρόνια ε, προβληματιζόμαστε. Κύριε Ερτούκ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προσθέσει κάτι. Η Ντεζεζίστε δεν είναι εδώ. Υπάρχει εδώ κάποιος από τον Ντεζεζίστε, όχι. Μάλιστα. Κύριε Ερτούκ, έχετε το λόγο. Ως εισηγητής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την DG Move και την DG Grow. Ήθελα να πω ότι δεν μπορεί κανείς ε, μόνο να φωνάζει από τον άμβονα της Εκκλησίας κατά των ε, αμαρτωλών. Ούτε και εγώ θέλω να πετροβολήσω την Κομισιόν. Έχω πληροφορίες εσωτερικές. που με κάνουν να πω ότι αυτές οι δύο γενικές κατευθύνσεις, ε, ευθύνσεις μάλλον που είναι σήμερα εδώ παρούσες, γνωρίζουν πολύ καλά το πρόβλημα. Η δυσκολία είναι ότι μέσα στην Επιτροπή κάποιες φορές είναι δυσκίνητοι οι μηχανισμοί και δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν ε, και τα, ε, πώς να οι επαφές ανάμεσα στις διάφορες διευθύνσεις. Εγώ δεν θέλω να στραφώ εναντίον ε, κάποιες από αυτές τις δύο διευθύνσεις που είναι παρούσες. Πάντως, η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μας θέλει σοβαρά να εμποδίσει αυτές τις απάτες που είναι εις βάρος των καταναλωτών. Και νομίζω πως πραγματικά υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην οδική ασφάλεια και ένα αυτοκίνητο το οποίο κυκλοφορεί και όπου έχει πειραγμένο κοντέρ. Αυτό θα πει ότι το σύστημα φρένου δεν είναι το ίδιο με ένα καινούριο αυτοκίνητο. Όταν ένα αυτοκίνητο έχει ήδη κάνει 120.000 χιλιόμετρα, ε, έχουμε ευθύνη. Έχει ευθύνη η αρμόδια γενική διεύθυνση που είναι εδώ. Δεν θέλει να δεν θέλει λοιπόν να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Βέβαια το κοινοβούλιο μας ε, έτσι δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο συνομοθέτης και ε, θέλω να επαναλάβω την πρόταση του συναδέλφου Βάντερ Κάμπ. Πιστεύω πως η πρόεδρος μας με τη στήριξη των συντονιστών θα πρέπει να στείλει επιστολή στον Τίμερμανς και μάλιστα να τον καλέσει εδώ, να μας εξηγήσει. Να μας πει ποιες είναι οι προθέσεις της Επιτροπής και για να δούμε αν θα καταφέρουμε να βρούμε το δίκαιο μας. Ο Τίμερ μας είναι έξυπνος άνθρωπος, όχι μόνο γιατί είναι σοσιαλδημοκράτης, αλλά και επειδή πιστεύω πως γνωρίζει τις μελέτες που αποδεικνύουν πόσο απαραίτητο είναι να δοθούν απαντήσεις. Φαντάζομαι ότι και ο Τίμερμανς έχει και άλλα επίγοντα θέματα που τον απασχολούν αυτή τη στιγμή. Όμως, εγώ δεν νομίζω πως ε, ωφελεί σε τίποτα το να συνεχίσουμε να ακούμε τους συναδέλφους της Κομισιόν, τους οποίους ε, Βεβαίω, καταλαβαίνουμε. Εγώ του εκφράζω την αλληλεγγύη μου γιατί γνωρίζουμε πως οι ευθύνε ε, δεν βαραίνουν τους δικούς τους ώμου, αλλά τους ώμου του ανώτερου επίπεδου. Ευχαριστώ και πάλι του συναδέλφου για την υποστήριξή τους λοιπόν που δείχνει ότι είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ερτούγκου. Σα διαβεβαιώνω ότι θα είναι στο θέμα στην ημερήσια μα διάταξη των συντονιστών που θα γίνει η συνεδρίαση αυτή στις 19 Μαρτίου για να δούμε τι θα κάνουμε για να ξυπνήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να έχουμε πια συγκεκριμένη απάντηση για αυτό το θέμα. Συνεχίζουμε τώρα με μια παρουσίαση για πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικά προγράμματα στον ε, μεταφορές και τον τουρισμό. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Κομισιόν ώστε να μας δείξει Ποια είναι η φάση στην οποία βρίσκονται τα πιλωτικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικέ δράσει, καθώ και τα αποτελέσματα των project που μόλι κλείσαν. Όπω ξέρετε, τα πιλωτικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικέ δράσει προτείνονται από το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο τη ζητήση δημοσιονομικής διαδικασία και σε λίγε εβδομάδε θα έρθει σε επαφή μαζί σα ή η Γραμματεία ώστε να διατυπώσετε νέε προτάσει σε σχέση με την δημοσιονομική διαδικασία του 19. Πιστεύω λοιπόν πως αυτή η παρουσίαση ε, είναι πολύ επικαιρή διότι πριν να υποβάλουμε νέε προτάσεις ε, καλό θα είναι να κάνουμε μια, δούμε μάλλον μια κατάσταση πρόοδου των όσων ήδη είχαν επιλεγεί. Δίνω το λόγο λοιπόν τώρα στην κυρία Κυρία Μόνα Μπόρχεντ, πού βρίσκεστε, μάλιστα. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Είμαι υπεύθυνη για τη μονάδα προγραμματισμού στη Γενική Διεύθυνση MOVE. Με χαρά είμαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω τα πιλωτικά και προπαρασκευαστικά προγράμματα στον τομέα των μεταφορών θα συμπληρώσει την παρουσίασή μου και η Γενική Διεύθυνση Growth για τον τουρισμό. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υποστηρίζει αυτού του είδους τα προγράμματα η ανάλυση η οποία οδηγεί στα προγράμματα αυτά παρέχει θα έλεγα χρήσιμες πληροφορίες και για τη γενικότερη πολιτική μας και για τις συζητήσεις που κάνουμε για τους τομείς αυτούς και σας ευχαριστώ για τούτο. Να μου επιτρέψετε να παρουσιάσω τα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει από το 2016 και μετά να σταθώ επίσης σε κάπως περισσότερες λεπτομέρειες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι οι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος ε, περιλαμβάνεται στην ετήσια ενδιάμεση έκθεση την οποία παρουσιάζουμε κατέτος τον μήνα Μάρτιο και μόλις καταθέσαμε στο τέλος Φεβρουαρίου την φετινή έκθεση. Σχετικά με το 2016 η Γενική Διευθύνση MOVE ασχολείται με τέσσερα, προπαρα... με πιλωτικά και δύο προπαρασκευαστικά προγράμματα. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ε, συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Τα προγράμματα αυτά έχουν αρχίσει τώρα να τρέχουν, να εξελίσσονται Έχουμε ολοκληρώσει όμως και κάποια προγράμματα όπως το σύστημα monitoring του ε, GNSS. Θα επανέλθω σε αυτό ε, και θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Ένα άλλο παράδειγμα όπου ο τομέας έχει ολοκληρώσει αν θέλετε τη μελέτη είναι τα ενιαία ευρωπαϊκά συστήματα και νοτομίες. Συνεχίζεται βέβαια η προσπάθεια σε, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα λεγόμενα πολυτροπικά ή multimodal προγράμματα. Οι δράσεις αυτές ξεκίνησαν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και θα συνεχιστούν. Από το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει με πέντε πιλωτικά προγράμματα, από τα οποία τα τρία έχουν παραταθεί μέχρι και το 2018. Βλέπετε τους μικρούς αστερίσκους ίσως στις παρουσιάσεις τους πίνακες. Για το 2017 λοιπόν υπήρξαν ρυθμίσεις για την χρηματοδότηση, έχουν ξεκινήσει οι ε, ε, διαγωνισμοί για τα προγράμματα αυτά. Θα έχουμε αποτελέσματα στο τέλος του χρόνου για το 2018 πέρα από τα τρία προγράμματα με τους αστερίσκους που προέρχονται από το 2017 έχουμε και τρία νέα πιλωτικά ε, στις ενδιάμεσες εκθέσεις μας. Ε, όλα αυτά αναφέρονται σε θέματα οδικής ασφάλειας, ε, ανθρώπινη συμπεριφορά και αυτόνομη ηλεκτρονική οδήγηση, Επίσης και αυτοματοποιημένα προγράμματα ευρωπαϊκά για τη μείωση των απατών στον τομέα των οδομετρητών ή των χιλιομετρητών. Ε, να σας δώσω κάποια επιπλέον παραδείγματα. για τα πιλωτικά του 2016 σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης που βασίζεται στο GNSS για τα εμπορικά βαρέα οχήματα. Εμείς αξιολογήσαμε λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα στα πλαίσια των προτάσεων βελτίωσης ε, ε, των ρυθμίσεων. Ε, κάναμε μια τεχνική ανάλυση κόστους-οφέλους για την επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας χρησιμοποιώντας τους ταχογράφους σαν βασικό στοιχείο. Ολοκληρώθηκε η μελέτη τον Ιούνιο του 2017 και μεταφέρθηκε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ανάλυση είναι θετική και δείχνει ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα ένα τέτοιο σύστημα στις οδικές μεταφορές, μια μείωση του παράνομου καμποτάζ επίσης και μείωση των χιλιόμετρων που διανύονται από τα φορτηγά. Ε, το επόμενο πρόγραμμα ξεκινά με πιλωτικό του 17 σχετικά με την, με την μεταφορά προσώπων περιορισμένης κινητικότητας. Στόχος είναι να καταλήξουμε σε ε, κάποιες προτάσεις ε, που θα προετοιμάζουν τους ταξιδιώτες αυτούς ε, για τις μετακινήσεις τους στην Ευρώπη. Θα ξεκινήσουμε μία μελέτη στα μέσα του 2018. Ε, καταρχάς ε, θα καταγράψουμε το σύνολο των μέσων που έχουμε και για μεσοπρόθεσμες μετακινήσεις ή και για πιο μεγάλης διάρκειας θα κάνουμε και ένα πιλωτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου οι ε, πληροφορίες που έχουν συλλεγεί στην πρώτη φάση θα εφαρμοστούν. Η τελική έκθεση αναμένεται στο τέλος του 2018 και νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτά θα μας βοηθήσουν να βρούμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για τη σωστή ενημέρωση των προσώπων περιορισμένης κινητικότητας και θα ληφθούν υπόψη σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το επόμενο παράδειγμα είναι ένα πιλωτικό του 2017 για ασφαλείς θέσεις στάθμευσης των φορτηγών. Είναι καρπός διαπραγματεύσεων που έγιναν για το πακέτο Mobility 1. Το πρόγραμμα αυτό έχει σαν στόχο την αξιολόγηση και τα κίνητρα που απαιτούν, των, κινδύ, των αναγκών μάλλον και των κινήτρων που απαιτούνται για την ασφαλή στάθμευση των φορτηγών. Οι μελέτες θα συνεχιστούν μέχρι τον Ιανουάριο του 2018, θα έχουμε όμως μία ενδιάμεση αξιολόγηση το Φεβρουάριο και θα οργανώσουμε μία σημαντική συνάντηση την 5η Νοεμβρίου επ' αυτού. Το επόμενο πρόγραμμα, πάντα του 2017, πιλωτικό για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Ε, θα παραταθεί και στα πλαίσια του 2018. Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας πρότασης για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό που να εμπνέεται από τις προτάσεις και τις δικές σας για τους λεγόμενους Trans-European Motorways of the Sky εμείς έχουμε μία συμφωνία με την ε, ΕΑΣΑ γύρω από αυτά και η πρόταση στις 9 Μαρτίου θα γίνει δεκτή επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο θα έρθουμε σε επαφή και σε διαβουλεύσεις με τους εμπλεκομένους και θα οργανώσουμε και εργαστήρια μελέτης. Θα ολοκληρώσουμε στο τέλος του χρόνου ε, την μελέτη και θα προχωρήσουμε στη συνέχεια στην φάση 2. Νομίζω ότι τα στοιχεία αυτής της μελέτης θα ληφθούν υπόψη για τις μελλοντικές εξελίξεις του πλαισίου του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Και τέλος το θέμα που συζητήσατε προηγουμένως για τις απάτες στον καταγραφέα των χιλιόμετρων, ταχογράφο. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει από το 17 και αναζητεί πιθανές λύσεις για την σωστή ανταλλαγή πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα ολοκληρωθεί στο τέλος της φετινής χρονιάς. Ε, νομίζω ότι ήδη θα έχουμε κάποια πρώτα στοιχεία τις επόμενες εβδομάδες και θα λάβουμε υπόψη και τη μελέτη τη δική σας. Η μελέτη όμως, συγγνώμη, θα παραταθεί το 2019. Νομίζω ότι αυτά είχα να πω στην παρούσα φάση, να, μετα... να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους από την Γενική Διεύθυνση Growth, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής Πολιτικής. Η κυρία Θανασοπούλου έχει το λόγο. Δεν έχει φτάσει όμως ακόμα η κυρία Θανασοπούλου. Alors, on revient sur la notion de tourisme Attendez, attendez. Λοιπόν, η ομιλήτρια που θα έπρεπε να είναι εδώ τώρα για τα θέματα του τουρισμού δεν είναι ακόμα παρούσα. Δυστυχώς γι' αυτήν θα ξεκινήσει η συζήτηση για το πρώτο κομμάτι σχετικά με τις μεταφορές. Και δίνω αμέσως το λόγο στον Βαντακάμπ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξηγήσεις τις οποίες μας έχει δώσει. Το δικό μου θέμα δεν είναι κάτι το οποίο έχει συμπεριληφθεί σε αυτά τα οποία ακούσαμε. Ε, θα ήθελα να εκφράσω μια άποψη για τους ασφαλείς χώρους στάθμευσης των φορτηγών. Είναι κάτι που ξεκίνησε από τον συνάδελφο Βαντάλεν ε, των ε, Ευρωπαίων Συντηρητικών. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας είπε ότι μέχρι τον Νοέμβριο ή 5 Νοεμβρίου θα γίνει μια συνάντηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα αυτό. Ελπίζω να έχουμε προχωρήσει στον τομέα του τριμερούς διαλόγου. Υπάρχει θέμα χρηματοδότησης αυτών των θέσεων στάθμευσης. Το πρόβλημα είναι σημαντικό. Πολλοί είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί γρήγορα αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν πριν ολοκληρωθεί μια τέτοια διαδικασία. το σχέδιο 34027703. για τον κύκλο ζωής των βιοκαυσίμων. Ε, τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι ε, πλήρη. Πάντως Ε, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τη μέθοδο VLTP. Ελπίζω να χρησιμοποιηθεί σαν πεδίο αναφοράς αντίθετα με την προηγούμενη μέθοδο του NDC. Λοιπόν, το προηγούμενο σύστημα με λίγα λόγια έχει ξεπεραστεί και θα πρέπει το νέο σύστημα να χρησιμοποιείται από εδώ και πέρα που θα περιλαμβάνει το σύνολο των εναλλακτικών καυσίμων και τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Θα υπάρχει δηλαδή ένα νέο ευρωπαϊκό ενεργειακό μίξ και θα περάσουμε στο αντίστοιχο μίξ που ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο που είναι διαφορετικό από αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για το προσδόκιμο ζωής του οχήματος το οποίο λαμβάνεται υπόψη. Αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί αρνητικά για τα εναλλακτικά καύσιμα και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα 200.000 χιλιόμετρα μπορεί να θεωρηθεί από ό,τι φαίνεται σαν στόχος αναφοράς, benchmark για όλα τα προγράμματα. Ευχαριστώ κύριε Βαντερκάμπ, ο κύριος Σέρτου Γκόχη. θέλω να ρωτήσω, άλλωστε ο Βαντερκάμπ ζήτησε πολλά πράγματα, Θέλω να ρωτήσω για το European 2. Ακούσαμε πριν και την παρουσίαση του ελεγκτικού συνεδρίου που είπε ότι θα πρέπει να γίνει περισσότερη επένδυση εκεί για το Single European Sky. Single European Sky. Περιλαμβάνεται και αυτό. Δεύτερο, ασφαλή θέση στάθμευσης. Τώρα που συζητούμε και για το European Mobility Package, πού γίνεται ακριβώς η έρευνα αναζητούνται best practices από άλλες χώρες μέλη, γίνονται έρευνες μόνο σε ορισμένες χώρες μέλη. Πώς, ποια είναι η προσέγγιση σε αυτό. Σήμερα Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάισνερ. Η κυρία Αιάλα Σέντερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες ε, την Επιτροπή. Και θα ήθελα να σχολιάσω το εξή. Πρώτο, είδα, ε, βλέπαμε ένα κατάλογο από μελέτες που ήδη έχουν γίνει, ολοκληρωθεί, και είδα εκεί τη μελέτη που αφορά την ελκυστικότητα του τομέα των μεταφορών. Όταν έχουν ε, ολοκληρωθεί λοιπόν οι μελέτες ε, πώς τις ξαναχρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας εργασία. Πώς τις ενσωματώνετε εκεί και θα ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Αντελή αν μπορούμε στην καθημερινή μας δουλειά να ενσωματώσουμε επίσης μια παρουσίαση αυτών των μελετών, γιατί ορισμένες εξ αυτών, όπως ας πούμε αυτό που αφορούσε την ελκυστικότητα του τομέα των μεταφορών για νέους ανθρώπους, για τις γυναίκες, μπορούσε ίσως όντως να ενδιαφέρει. να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα στο μέλλον. Μετά υπάρχει μια άλλη μελέτη ε, που δεν την είδα εδώ στο κατάλογο, αλλά μάλλον επειδή δεν πρόλαβα και αφορά την ανθρώπινη συμπεριφορά στη διάρκεια της αυτόνομης οδήγησης. Και θέλω να ξέρω τι γίνεται με αυτή τη μελέτη, γιατί δεν την είδα στον κατάλογο. Μπορεί εγώ να μην πρόλαβα να το δω, αλλά θέλω να ξέρω πού βρίσκεται αυτή η μελέτη και πώς μπορεί κανείς να, να, τη δει ε, ολοκληρωμένη όσο γίνεται πιο σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Λύρη. DG Grow-nak a képviselőit, turizmus kapcsán tudjunk egyeztetni, de hát ugye... Εδώ περιμένουμε την εκπρόσωπο της Digigrowth Growth για το θέμα του τουρισμού. Αλλά εγώ έχω ένα γενικότερο ερώτημα, το οποίο θα ήθελα να θέσω υπόψη των μελών της Επιτροπής Μεταφορών και βεβαίως και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δαπανά περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για διάφορα πιλωτικά προγράμματα για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω τι γίνεται σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που βλέπω όμως εδώ και που παρατηρώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίζεται τα χρήματα αυτά. Καλά βεβαίως τα έχουμε θέσει τη διάθεσή της εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο, αλλά εμείς οι ευρωβουλευτές που έχουμε δουλέψει τόσο πολύ για να εξασφαλίσουμε τα κονδύλια αυτά, βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέναντί μας να μην θεωρεί ότι είναι υποχρεωμένη να λογοδοτήσει. Αυτό δεν είναι σωστό. Γι' αυτό χαίρομαι που τέθηκε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη, διότι πρέπει να πούμε μια και καλή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα πιλωτικά αυτά προγράμματα υπάρχουν και εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς ακριβώς επειδή ορισμένοι ευρωβουλευτές έχουν εργαστεί σκληρά για να προωθήσουν συγκεκριμένα οράματα. και έχουν εξασφαλίσει τα σχετικά κονδύλια. Τα τελευταία χρόνια 11 περίπου εκατομμύρια ευρώ έχουμε κατορθώσει να εξασφαλίσουμε για τον τουρισμό. Και εδώ οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστήσεις μου στην Επιτροπή Μεταφορών, η οποία μας εστήριξε στον αγώνα αυτόν. Όμως δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα που έχουν πάει τα χρήματα αυτά. Και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε έτσι, αυτό ε, θα απογοητεύσει τους ευρωβουλευτές ενώ οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν είναι εκλεγμένοι και επομένως δεν λογοδοτούν σε κανένα ψηφοφόρο, αυτοί λοιπόν οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εργάζονται ως υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαχειρίζουν τα χρήματα αυτά χωρίς να μαθαίνουμε εμείς τους σκοπούς για τους οποίους δαπανώνται. υπάρχουν συναδελφοί μου ε, που συνεργάζονται μαζί μας, αλλά το πρόβλημα που εντοπίζω είναι συστημικό. Διότι μας απαντούν κάθε φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπόχρεη να λογοδοτήσει. Δεν είναι υποχρεωμένη να εξηγεί στους ευρωβουλευτές τι γίνεται με τα πιλωτικά προγράμματα τα οποία εμείς οραματιστήκαμε και για τα οποία εμείς εξασφαλίσαμε τα κονδύλια. Και αυτό θα σας το βεβαιώσουν και άλλοι συνάδελφοι ευρωβουλευτές. Θέλω λοιπόν να ζητήσω το εξή προς το συμφέρον της σωστής εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να απαιτούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λογοδοτεί ενώπιόν μας για το πού ξοδεύει τα χρήματα αυτά. Η δε ευρωβουλευτές οι οποίοι είχαν την αρχική ιδέα για το συγκεκριμένο πιλωτικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι παρόντες κατά τη ε, διαδικασία αυτή λογοδοσίας. Εμείς έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να ενισχύσουμε νέους ανέργους, για να φτιάξουμε προγράμματα επανεκπαίδευσης, ώστε τα πρόσωπα αυτά να μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα τουρισμού. Γνωρίζετε όλοι ότι στην Ανατολική Ευρώπη η αγορά εργασίας είναι πολύ διαφορετική από την, ας στο Λονδίνο ή σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις της Δυτικής Ευρώπης. Μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε κάποια κονδύλια και είδα μετά από ένα εξάμεινο ότι το πρόγραμμα λειτουργήσε υπό άλλο όνομα. και ανατέθηκε στην μια κοινοπραξία η διαχείρισή του που δεν είχε απολύτως καμιά σχέση με την Ανατολική Ευρώπη. Ενώ ο σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να ενισχύσει τέτοιες προσπάθειες στην Ανατολική Ευρώπη. Ζητώ τη συνεργασία των συναδέλφων μου λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας, τις οποίες στηρίζουμε. Πρέπει και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξέρουμε πού πάνε αυτά τα χρήματα και για αυτό το θέμα της ε, ε, χρηματοδότησης και της διαφάνειας. Εγώ έχω δύο-τρεις ερωτήσεις ε, να σας κάνω, αν μου επιτρέπετε. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα για τον οδομετρητή. Δεν είμαστε όμως ε, ευθυγραμμισμένοι γιατί η μελέτη θα ολοκληρωθεί όταν θα έχουμε ήδη προχωρήσει την έκθεση πρωτοβουλίας και θα έχουμε... Ποια είναι η μέθοδος για την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσουμε ώστε για να μην είναι υπεπαλαιωμένη μόλις ολοκληρωθεί αυτή η έκθεση για τον, για τον οδομετρητή Δηλαδή δεν χρειάζεται να δαπανίσουμε 300.000 ε, ευρώ για αυτή τη μελέτη, αυτή τη εφού δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε τα πορίσματά της τελικά. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερο, ε, όλα αυτά τα project τα οποία έχετε αναφέρει ε, και όντω αφορούν την κινητικότητα, πώς θα κάνουμε όμως σήμερα ώστε και αύριο, γιατί ο κύριος Γλύρη λέει πρέπει αυτά τα project να τα παρακολουθούμε. Πώς λοιπόν αύριο μεθαύριο αυτά τα πιλωτικά προγράμματα θα μπορέσουν να γενικευθούν. Αν υπάρχουν καλά μέτρα, καλά μέτρα θετικά, πώς λοιπόν αυτά τα πιλωτικά θα μετατραπούν σε πραγματικές δημόσιες πολιτικές και να μην είναι μόνο ε, μικρά προγραμματάκια που αύριο μεθαύριο δεν θα, θα έχουν ξεχαστεί ενώ λειτουργούν Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στην κυρία Μόνα Μπόκλαντ για να απαντήσει σε αυτά όλα και να δώσω και σύντομα το λόγο στην Κομισιόν για την πτυχή του τουρισμού. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. Ε, δύο λόγια για να απαντήσουμε στα ερωτήματα για τους ασφαλείς χώρους στάθμευσης για τα βαρέα οχήματα. Υπάρχουν διάφορα project και όπως είπε ο κ. Ε, Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι οι χώροι στάθμευσης είναι ασφαλείς και ασφαλισμένοι. Τι είδους μέτρα πρέπει να λάβουμε και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε πού θα τοποθετηθούν αυτοί οι χώροι στάθμισης και πόσοι θα χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες που υπάρχουν. Ποιο είναι ένα σωστό πλαίσιο για να δοθούν κίνητρα στους ε, ενδιαφερόμενους. Αυτό είναι κάτι που θα τοποθετηθουν αυτοι οι χωροι σταθμευσης και ποσοι θα χρειαζονται για να ανταποκριθουν στις αναγκες που υπαρχουν ποιο ειναι ενα σωστο πλαισιο για να δοθουν κινητρα στους ενδιαφερομενους αυτο ειναι κατι που θα γινει μέσα από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο συμπληρώνει και το κομμάτι της χρηματοδότησης ε, όπου υπό αυτό το πρόγραμμα έχουμε δεσμεύσεις ε, για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και να δημιουργήσουμε ασφαλείς χώρους στάθμευσης σε πολλά χιλιόμετρα δρόμο. Αυτό υπάρχει ήδη, τα κατημέλη ήδη μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ώστε να μπορέσουν να κατασκευάσουν αυτό το δίκτυο που χρειάζεται. Για τα θέματα για τον κύκλο ζωής των ηλεκτρικών οχημάτων Θα πρέπει αυτό να το παραπέμψω στους ειδικού μας στη Γενική Διεύθυνση και να σας ενημερώσω διμερώς αν θέλατε αργότερα. Για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, η ερώτηση ήταν αν θα λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα των συμπερασμάτων του ελεκτικού συνεδρίου. Βεβαίω τα πιλωτικά project αυτά είναι έτσι ε, φτιαγμένα ώστε να μπορούμε να βασιστούμε σε όλες τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας και φυσικά και θα τις ε, προσέξουμε. Την ανάγκη για επενδύσεις, ναι, και γι' αυτό το λόγο αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα είναι πολύ επίκαιρο. Θα μας επιτρέψει να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε με τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες. Αυτό μας δείχνει ήδη πόσο χρειάζεται να επενδύσουμε σε αυτό το τομέα. Τώρα, ε, θέματα για το τι γίνεται μόλις ολοκληρωθεί κάθε μελέτη. Είναι πολύ καλή ερώτηση και εδώ η πρακτική ε, διαφέρει. Ε, ήδη, ας πούμε, στην προετοιμασία κάποιων project το συζητάμε εδώ με το Κοινοβούλιο, όμως όταν έχει ολοκληρωθεί μια μελέτη, φιλάσετε, φυλάσσετε, ε, σας ενημερώνουμε σχετικά και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας εάν επιθυμείτε κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια ε, μελέτη. Τώρα, από τη δικιά μας πλευρά χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές. Είμαστε μια κομισιόν που λειτουργεί με βάση τα στοιχεία. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία και τις αναλύσεις κάθε φορά, ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε για να... και να προτείνουμε λύσεις, αλλά βεβαίως μπορούμε να μελετάμε και από κοινού τα ίδια έγγραφα. Τώρα, για την αυτόνομη οδήγηση. Αυτό είναι κομμάτι των πιλωτικών προγραμμάτων για το 2018 αυτά που είδατε στις διαφάνειες. Αυτά που τώρα αρχίζουμε και τώρα λαμβάνονται οι αποφάσεις περί χρηματοδότησής τους θα τα ε, δείτε αργότερα. Για την μελέτη που είπατε, το διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση είναι πρόταση του 2018 ε, και βεβαίως δεν θα το προχωρήσουμε. Ε, θα θα, θέλουμε να αναλύσουμε και να εκτιμήσουμε το θέμα, αλλά βεβαίως και σημειώνουμε ότι σας δεν θα σας χρησιμεύσει. Και πάλι, και ναι, νομίζω απάντησα στο θέμα της ε, λογοδοσίας, ίσως καλύτερη χρήση και ανταλλαγή των πορισμάτων, των πιλωτικών προγραμμάτων. Πέρα αυτού είμαστε, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για το σύνολο των απαντήσεών σας και τώρα στρέφομαι προς τον συναδελφό σας. Τι συναδελφό σας που ασχολείται με ε, το, ε, την πτυχή του τουρισμού. Κυρία Άννα Αθανασοπούλου. Ωραία το είπα, λέει η Πρόεδρος. Ναι. Ε, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, τέλεια το είπατε. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε μια γενική εικόνα για την εφαρμογή των πιλωτικών προγραμμάτων περί τουρισμού και των προπαρασκευαστικών δράσεων και ζητώ συγγνώμη που άργησα και έχασα την αρχή πήγατε λίγο πιο γρήγορα στη μερική διάταξη. Ζητώ συγγνώμη. Και πάλι η σημερινή μα εισήγηση συμπληρώνει τι γραπτέ πληροφορίε που ε, λάβατε, ε, που λαμβάνετε μάλλον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο τη ετήσια ε, διάμεση έκθεση για την εφαρμογή των πιλωτικών προγραμμάτων και προπαρασκευαστικών δράσεων και τα έγγραφα εργασία που συνοδεύουν το σχέδιο προπολογισμού για τον επόμενο χρόνο. Με βάση αυτέ τι πληροφορίε που ήδη φτάνουν τακτικά στο Ευρωκοινοβούλιο, θα σας παρουσιάσουμε σύντομα ένα περίγραμμα των αποτελεσμάτων των δράσεων που έχουμε εφαρμόσει μέσω, μέσω αυτών των, τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Για την περίοδο 2015 με 18 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει νέα πιλωτικά project και προπαρασκευαστικές δράσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό με σύνολο προϋπολογισμό 11,1 δις. Ε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ευρωκοινοβούλιο που πρότεινε αυτά τα project και για το ενδιαφέρον που δείχνει για τον τομέα του τουρισμού. Θα ξεκινήσω με το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα αύξηση των, ε, των, θέσεων, ποιοτικών θέσεων εργασία και των μαθητιών στον τουριστικό τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι γνωστό και ως Youth on the Spot ε, και προτάθηκε με 500.000 ευρώ υπό τον προπολογισμό του 2016. Αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα εστιάζει σε τουριστικές αδιαδρομίες να βελτιώσει την ελκυστικότητα των ε, θέσεων απασχόληση στον τουρισμό και να βελτιώσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών του το τομέα του τουρισμού. Μόνο έχουμε έξι υποτομείς, δηλαδή στέγαση, γαστρονομία, ε, διαχείριση προορισμού, ε, τουρ, ε, ψηφιακές υπηρεσίες και καινοτομία. Ενώ το project εστίασε σε 8 κρατη τελικά τα αποτελέσματά του, τα πορίσματά του μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλα και ελπίζουμε πως μέσω της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε θα δούμε ωφέλη και σε άλλα κράτη-μέλη. Τώρα, ε, τα κύρια προϊόντα αυτού του project είναι ε, υλικό επικοινωνίας και πρόθεσης υπό τη μορφή βίντεο και φυλαδίων μια πλατφόρμα με πακέτα ε, ε, EU Learning για, για τους αναζητώντες εργασία, εργαλειοθήκες το ένα για τα μονοπάτια για τις τουριστικές σταδιοδρομίες και το δεύτερο για τις ευρωπαϊκές θέσεις και τη ε, εξέβρεση των ευκαιριών στον τομέα των ε, τουριστικό. Οχτώ σεμινάρια με τρόπους ε, αναζήτησης θέσεων. Επίσης, σε άλλα σεμινάρια για την αναζήτηση των κενών στις δεξιότητες και άλλα σεμινάρια όσον αφορά την επικοινωνία και τη διάδοση των υπαρχουσών θέσεων στον τομέα του τουρισμού. Το project αυτό απασχόλησε 5.000 κόσμο μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης. Ε, κύριοι βουλευτές, θα έχω την ευκαιρία να ακούσουν περισσότερα όσον αφορά τα αποτελέσματα αυτού του πιλωτικού προγράμματος στι 2 Απριλίου, όπου ο αρχηγό του προγράμματο θα κάνει μια εκτεταμένη παρουσίαση στο Ευρωκοινοβούλιο. Επίσης θα καταλανοήσετε ότι υπάρχει και μια συσχέτιση ανάμεσα στην συνέχιση της πολιτικής, των στόχων και των πορισμάτων αυτού του project και το χάρτη για την ε, συνεργα... το... διατομιακή συνεργασία στον τουρισμό είναι ένα project υπό το έρασμος ΣΥΝ, ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε κενά στις δεξιότητες και να παρουσιάσουμε πιο στοχευμένες δεξιότητες για τον τουριστικό τομέα μέσω και μακροπρόθεσμα. Να συνοψίσω τώρα τα συμπεράσματα, τα αποτελέσματα μάλλον της προπαρασκευαστικής δράσης ε, για τα ε, διακρατικά τουριστικά προϊόντα. Αυτή η προπαρασκευαστική προπαρασκευαστική δράση ε, πήρε 3 εκατομμύρια ευρώ. Η δράση αυτή μας επέτρεψε να ενισχύσουμε τη συνεργασία με την UNESCO, αναπτύσσοντας το πρώτο διαδρομές παγκόσμιες κληρονομιάς μέσα στην Ένωση. Αυτές οι διαδρομές ε, ε, αποτελούνται από αυτόματες διευρωπαϊκές διαδρομές που συνδέουν 24 πολύ γνωστές πολιτιστικές κληρονομιές της UNESCO και κάποιες λιγότερο γνωστές τα τέσσερα θέματα είναι η Βασιλική Ευρώπη, η Ρωμαντική Ευρώπη, Αρχαία Ευρώπη και η Υπόγεια Ευρώπη. Και ε, η προώθηση αυτών των διαδρομών έχει ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία με το National Geographic και θα συνεχιστεί στη δεύτερη φάση της προπαρασκευαστικής δράσης που έχει ξεκινήσει τον Ιανουάριο φέτος και θα συνεχιστεί για 18 μήνες. Μέχρι στιγμής ε, τα στόχοι είναι η δουλειά ε, για την δημιουργία δυνατοτήτων και για εργαλειοθήκες, εργαλεία μάλλον και σεμινάριο, μια βελτιστοποιημένη πλατφόρμα όπου προωθούνται αυτές οι διαδρομές και στοχευμένες δραστηριότητες πρόθεσης συνεργασία με το National Geographic, όπως ήδη σας είπα. Um, uh, η προσπάθειά μας είναι να προωθήσουμε αυτές τις διαδρομές περισσότερο μέσα στο 2018 και μέχρι και τα μέσα του 2019 να αυξηθεί η ορατότητά τους με ιδιαίτερη ε, ε, ε, στόχο τις μακρινές αγορές όπως η Κίνα. Μάλιστα φέτος είναι και το έτος ε, τουρισμού Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα, αλλά και με τη Βόρεια Αμερική θέλουμε να διαδοθούν. Τα αποτελέσματα αυτά θα τα δείτε στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων και δυνατοτήτων προώθησης στο πλέτο του έτους τουρισμού Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς, εφόσον υπάρχει συσχέτιση με την πολιτιστική κληρονομιά και βέβαια με την κοινή πλατφόρμα Πρόθεση, μια νέα πρωτοβουλία που εφαρμόζουμε από κοινού μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ταξιδίων και που θα σας εξηγήσω αργότερα στην εισηγήσή μου. Πέρα από τις διαδικασίες πρόθεση σε σχέση με αυτές τις τέσσερις διαδρομές, Στόχο είναι να διευκολύνουμε τη συνεργασία ανάμεσα στην κληρονομιά και στι ε, αρχές ε, διαχείριση στον, τοπικές αρχές μάλλον στον προορισμό και ιδιαίτερα όσον αφορά ε, την πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Να στραφώ τώρα σε ένα άλλο πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά διαφορετικό θέμα. Ο τίτλος είναι ο ε, παγκόσμιος τουρισμός για ε, παγκόσμιος τουρισμός με 700.000 ευρώ χρηματοδοτήθηκε και το Κοινοβούλιο χρειάστηκε να το συνεχίσει ως προπαρασκευαστική δράση με ένα επιπλέον προπολογισμό 1,1 ε, εκατομμύριο. Λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού που είχαμε στην πρώτη φάση και του στόχου που έθεσε ο στο Κοινοβούλιο, αποφασίσαμε να στοχεύσουμε σε τρεις, σε τρεις πτυχές. Να δημιουργήσουμε με περισσότερε ευκαιρίε ανάμεσα στι ευρωπαϊκέ και τι κινέζικε εταιρείε, να γνωρίσουμε το προφίλ των Κινέζων ε, ταξιδιωτών, ε, καθώ και να ετοιμαστούμε για σε σχέση με την Κίνα. και αυτά ε, συντονίζονται με τους ευρύτερους στόχους, ε, όπως είπαμε, ε, για το έτος τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Μέσα από αυτό το πιλωτικό project έχουμε διάφορες εκθέσεις κάνει, υπάρχουν δε και στα διάφορα website που χρησιμοποιούνται από τους φορείς του τουρισμού. Κάναμε διάφορα σεμινάρια μέσω του διαδικτύου, αλλά και workshops στην το ένα στη Σανγκάη και το άλλο στο Λονδίνο. Και έχουμε και διάφορα ταξίδια ε, εξοικείωση για τους Κινέζους ε, operators. Βεβαίως εδώ θα ε, δούμε πιο απτά τα αποτελέσματα στη διάρκεια της ημερίδας για το πιλωτικό πρόγραμμα ε, τουρισμός που γεφυρώνει τις αποστάσεις. Έχουμε ακόμα ένα project για να προωθήσουμε την Ευρώπη ως προορισμό, τουριστικό προορισμό, όπου είχαμε συνολικό προπολογισμό 1,5 εκατομμύρια ευρώ και για να μπορέσουμε εδώ να μοχλεύσουμε περισσότερα ε, με βάση τον αρχικό προπολογισμό που μας έδωσε το Κοινοβουλίο, σωρέψαμε αυτόν τον προπολογισμό με τον κανονικό μας προπολογισμό ε, υπό το κόσμο και, και επιπλέον κονδύλια τα οποία παίρνουμε από το Ευρωπαϊκό Κονδύλιο Ναυτιλίας. Έτσι λοιπόν μπορέσαμε να φτιάξουμε μια κοινή πλατφόρμα προώθησης για την Ευρώπη ως προορισμό και αυτό εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχο έχει να αναπτύξει και να διαδώσει ευρωπαϊκές δραστηριότητες για ευρωπαϊκά και διευρωπαϊκά προϊόντα και σε στοχευμένες τρίτες χώρες. Η καινοτομία είναι όχι ότι έχουμε συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών, των μάνατζερ, αλλά έχουμε και ιδιωτικές εταιρείες και operators. Ελπίζουμε στα πλαίσια αυτών των προπαρασκευαστικών δράσεων να προχωρήσουμε. Ζητήσαμε και μία προπαρασκευαστική από εσά για φέτος για την προώθηση των πολιτιστικών θησαυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε επίσης και για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Εφιούς Τουρισμού. Ξεκίνησε ήδη η προσπάθεια από τον Ιανουάριο, η δράση. Έγκυται στην επιλογή δύο πόλεων ως Ευρωπαϊκών Πρωτεύουσων από το 2019 Ευρωπαϊκών Πρωτεύουσων του Τουρισμού βασική ιδέα είναι να αναγνωρίσουμε στις πόλεις τις προσπάθειες που κάνουν για ευφυΐες τομείς τουρισμού, ε, συστηματικότητα, προσβασιμότητα, ε, πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά. Ζητάμε την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προπαρασκευαστική της συγκεκριμένη δράσης Ελπίζουμε να πάρετε μέρος και στην Επιτροπή Επιλογής. Προβλέπετε μια πρώτη συνάντηση τον Νοέμβριο του 2018. Βλέπετε, Πρόεδρε, ότι κάνουμε προσπάθειες έτσι ώστε να προωθήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τις δράσεις μας. Σημεριζόμεθα μαζί σας την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προορισμού Ευρώπη και ελπίζουμε να συνεχίσουμε την ε, επιδίωξη επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Να πω ότι είναι πολύ περίπλοκο για μας να παρακολουθήσουμε ε, χωρίς ε, διαφάνειες αυτά τα οποία μας είπατε ε, στα πλαίσια της παρουσίασης της κυρίας Μπόρκλουντ είδαμε, βάση περιπτώσει, συγκεκριμένα στοιχεία γραπτά. Είδαμε επίσης συγκεκριμένες προτάσεις, ενώ η δική σας παρουσίαση είναι χωρίς διαφάνειες και δεν παρακολουθούμε μερικές φορές αυτά τα οποία λέτε. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα συζητήσουμε τα πιλωτικά προγράμματα μαζί, Παρακαλώ να στείλετε νωρίτερα στην γραμματεία μας λίγο πριν τα στοιχεία γραπτά. Και θα σας δώσω το λόγο μετά, εφόσον κάποιοι συνάδελφοι έχουν να κάνουν ερωτήσεις για τον τουρισμό. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, ο κύριος Βαντερκάμπ για λίγα λεπτά παρακαλώ. Βιμ Βαντερκάμπ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια σύντομη ερώτηση, μάλλον καλύτερα μια σύντομη παρατήρηση. Οι ειδικοί στα θέματα του τουρισμού οι συνάδελφοί μας εννοώ δεν είναι παρόντες. Πάντως την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια σημαντική συζήτηση για τον τουρισμό και την Κίνα. Και εγώ έθεσα ένα ερώτημα σχετικά με την αμοιβαιότητα. Ένας Κινέζος τουρίστας είναι διατεθειμένος να επισκεφθεί την Ευρώπη αλλά θα πρέπει να εμείνουμε λίγο στην εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας. Ε, μπορούν ας πούμε οι ε, ξεναγοί, οι Ευρωπαίοι να πάνε στην Κίνα και να εργαστούν εκεί. Μία απλή ερώτηση ήταν αυτή, τίποτα άλλο. Ε, ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Η Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ελπίζω να πήραμε λοιπόν, πήραμε ικανοποιητική απάντηση από τη Γενική Διεύθυνση MOVE και θα θέλαμε αντίστοιχες απαντήσεις και για τα πιλωτικά προγράμματα τα συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα για την προπαρασκευαστική βάση, δράση συγγνώμη, τριετούς διάρκειας ε, πρωτοβουλία καλύψω σχετικά με την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών για όλα τα επίπεδα, τα κοινωνικά δηλαδή και ηλικιωμένου και μεγάλες οικογένειες και κατηγορίες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να χρησιμοποιήσουν ε, τις ε, δυνατότητες τουρισμού. Ξέρουμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και είδαμε ότι ένας από τους δείκτες είναι ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή και η εργατική τάξη επίσης η οποία εθίγει κυρίως και για τις κατηγορίες αυτές τις ε, κοινωνικές οι διακοπές ήταν μια κοινωνική κατάκτηση για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, αλλά δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ισχύσει πλέον λόγω της ανεργίας για πολλούς και πολλοί από αυτούς έχουν αποκλειστεί από τέτοιου είδους δραστηριότητες. Γνωρίζει αυτή την προπαρασκευαστική δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα τη υπόψη της και με ποιο τρόπο. Εμείς περιμέναμε ένα ευρύτερο πλαίσιο για τέτοιου είδους προσπάθειες διευκόλυνσης ε, στις πρόσβασης σε τουριστικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ. Τελευταίος ομιλητής. Και η Επιτροπή θα έχει δύο λεπτά για να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. απευθύνομαι στην Άννα, η οποία ήταν απούσα προηγουμένω όταν τοποθετήθηκα, γιατί αρχίσαμε βέβαια την συζήτηση νωρίτερα. Θα διαβιβάσω όμως ε, το κείμενο της ομιλίας μου που εξεφώνησα προηγουμένως στην Άννα. Διότι περί τίνος επρόκειτο. Με λίγα λόγια αυτό που είπα είναι ότι τα κονδύλια τα οποία συλλέγονται με δική μας φροντίδα δαπανώνται για διάφορες εκδηλώσεις, συναντήσεις και ούτω καθεξής. Εμείς ωστόσο με τα χρήματα αυτά θέλουμε να διεξαγάγουμε πολιτική υπέρ της Ευρώπης. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει σφάλμα κάποιων ευρωβουλευτών ή κάποιων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι πάσχει το σύστημα. Προτείνω λοιπόν οι συντονιστές της Επιτροπής μας να εγκύψουν στο θέμα και θα πρέπει να ρωτήσουμε, να υποβάλουμε ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την ηγεσία του Πρόεδρου του κ. Γιούνκερ να μας εξηγήσουν πού πάνε τα χρήματα αυτά. Αυτό δεν είναι υπόθεση ειδικά των σοσιαλδημοκρατών, δεν ασχολούμαστε εμείς ειδικά με αυτό. Γι' αυτό συνιστώ να αναλάβουν πρωτοβουλία οι συντονιστές. Επαναλαμβάνω ότι δεν ευθύνονται κάποιες μονάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει σφάλμα στο ίδιο το σύστημα, το οποίο δεν επιτρέπει να προχωρήσουμε ικανοποιητικά. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών νομίζω η μερίσια διάταξη θα είναι αρκετά φορτωμένη. Όμως θα παρακαλέσω τώρα την κυρία Άννα Άθανασοπούλου να απαντήσει στο σύνολο των ερωτήσεων που έθεσαν οι συνάδελφοί μου και την παρακαλώ να περιοριστεί σε δύο λεπτά. Ορίστε κυρία μου, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά την αμοιβαιότητα των δράσεων, αμοιβαιότητα με την Κίνα, όπως είπα τα δύο matchmaking event που οργανώσαμε για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κίνα, το ένα έγινε, μία εκδήλωση έγινε στην Σανγκάη και η άλλη στο Λονδίνο. Και μέσα στο 2018, που είναι έτος κινέζικου τουρισμού, οργανώνουμε εκδηλώσεις για λογαριασμό επιχειρήσεων, όχι μόνο ε, δηλαδή, για να τις επισκεφτούν επιχειρήσεις, και εδώ στην Ευρώπη, αλλά και στην Κίνα, Σανγκάη και Μακάο. Πρόκειται λοιπόν για αμοιβότητα. Να μου επιτρέψετε να παραδώσω το μικρόφωνο στη συνάδελφό μου για να μπορέσει να απαντήσει στις ερωτήσεις για την προπαρασκευαστική δράση καλυψώ. Πριν το κάνω αυτό, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε διαβιβάσει μία σύντομη παρουσίαση PowerPoint στη γραμματεία σας. Ίσως ε, για κάποιο λόγο να ε, χάθηκε και να μην εμφανίστηκε στις οθόνες. Δεύτερο, στην παρουσίαση ίσως να μην ήταν σαφές, επιτρέψτε μου όμως να το επαναλάβω. Η προσπάθειά μας είναι να διασυνδέσουμε τα αποτελέσματα των project αυτών με πολιτικές οι οποίες κινούνται ούτε ούτε ή άλλως, είτε για δεξιότητες στον τομέα του τουρισμού, είτε για την προώθηση της ε, Ευρώπης ως ε, τουριστικό προορισμό ή για άλλα θέματα τουρισμού. Επιτρέψτε μου να δώσω το μικρόφωνο στη συνάδελφό μου. Κυρία Αγιάδα Σέντερ, γνωρίζω ότι ενδιαφέρεστε πολύ για τη συγκεκριμένη αυτή προπαρασκευαστική δράση και συνεχίσαμε και μετά από το τέλος της. Υπάρχει μάλιστα ένα σχέδιο δράσεως το οποίο έχει συνταχθεί με την βοήθεια εμπειρογνωμόνων του τομέα και μπορούμε να σας το διαβάσουμε. Έχουμε και διασύνδεση με την DG Connect για θέματα active aging για να δημιουργήσουμε συνεργασίες με αυτούς και έχουμε δώσει και ιδιαίτερη έμφαση σε προσκλήσεις ενδιαφέροντος στα πλαίσια της δράσης κόσμε. Και βέβαια για να διαφοροποιηθεί η προσφορά και να απευθυνθεί σε πλήρωνες ομάδες είτε ηλικιωμένων ατόμων είτε νεολαιών κλπ. Και δείχνουμε ιδιαίτερα, ε, ιδιαίτερη ευαισθησία σε όλες τις δράσεις μας για την λεγόμενη seasonality που γνωρίζουμε ότι είναι πρόκληση για όλο τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ κυρίες για τις απαντήσεις που δώσατε. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ειδωθούμε ξανά σύντομα και με περισσότερες πληροφορίες. Διότι το θέμα του τουρισμού είναι κέρια σημασίας στην δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αγαπητέ Βάντε Κάμπ, αν δεν έχετε διάφορα, δεν έχετε κανένα διάφορο. Καλά λοιπόν τότε. Η επόμενη συνάντησή μας θα διεξαχθεί την Δευτέρα 19 Μαρτίου από τις 3 και μετά. Σας περιμένω πολυάριθμους και πολυαριθμούς. Καλή εβδομάδα εδώ στην Ευρωβουλή.